Ας ξεκινήσουμε τις συνεδρίες της Επιτροπής. Έχουμε λιγότερο από μία ώρα στη διάθεσή μας για το σημείο 16 της ημερησίας διάταξης, τροποποίηση του κανονισμού 1234 του 2007 του Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Η συγγετής είναι ο κύριος Τζέμις Νίκολσον. Είναι σημαντικό η πρόταση της Επιτροπής να εξεταστεί εδώ στη δική Επιτροπή και να έχουμε συνεισφορά από όλες τις ομάδες. Ευχαριστώ και τον ε, Διευθυντή Ούλκερ, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρευρίσκεται εδώ σήμερα. Έτσι λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως και να δώσω το λόγο στον James για να κάνει μια εισαγωγή και κατόπιν φυσικά θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Uh, thank you Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξεκινώντας, ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν στην, θέσπιση, στην εκπόνηση αυτής της έκθεση, Φαντάζομαι ότι έχετε ήδη δει το κείμενο το σχέδιο για το πακέτο το σχετικό με τα χαρακτοκομικά. Ε, το είχαμε στα αγγλικά αρχικά, αλλά φαντάζομαι ότι μεταξύ είναι έτοιμο σε όλε τι γλώσσε. Θα ήθελα μέρα πολύ σύντομα να εξηγήσω τι κύριε τροπολογίε τη εκθεσή μου για να ακούσω τι απόψει των συναδέλφων, σχεδόν και των λοιπόν βουλευτών ε, για τα θέματα αυτά. Για να τα λάβω υπόψη μου για να τις λάβω υπόψη μου. Είχαμε λοιπόν κάνει τη συζήτηση με παρουσία και πολλών εκπροσώπων ε, και ενδιαφερομένων φορέων. Ε, φυσικά υπάρχει απόκληση απόψεων σε αρκετού τομεί, κυρίω μεταξύ εκείνων οι οποίοι έχουν, ε, εκπροσωπούν την ε, κατεργασία του γάλακτος και εκείνους που εκπροσωπούν τον παραγωγό ή τους παρατησινούς παραγωγών. Προσπαθώ λοιπόν εγώ με τις προτάσεις μου να ισορροπήσω τις διαφορετικές απόψεις θα μου πείτε εσείς αν τα κατάφερα. Σχετικά καταρχάς με τις ε, συμβάσεις και τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις συμβάσεις που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπου ξεκινάμε με την ε, καταβαλ... καταβληθισμένη τιμή. Ε, έχω ξεκινήσει εγώ με μια πρόταση για ρήτρε διαπραγμάτευσης όπου δεν θα είναι υποχρεωμένος ο παραγωγός να καταθέτει, να παραδίδει μάλλον ολόκληρη του την παραγωγή 100% σε έναν μόνο ε, εκπρόσωπο της, ε, του κλάδου της κατεργασίας. Μεγαλύτερη ευελιξία λοιπόν. Επίσης, σημειώνω ότι θα πρέπει σε επίπεδο κράτους μέλους να είναι μόνο εθελοντικές, υποχρεωτικά εθελοντικές αυτές οι συμβάσεις, ε, ακόμη και σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν έχει κάνει την επιλογή του opt στο σύστημα. Συμβάσει λοιπόν με τους παραγόγους θα υπάγονται στις ίδιες συνθήκες που προσδιορίζονται στην πρότασή μας. Όσον αφορά τους, ε, τη διαπραγματευτική ισχύ, θα δείτε ότι τα ποσοστά τα έχω μειώσει στο 20% το 23% ε, περιμένω να δω βέβαια τι τροπολογίε των συναδέλφων που θα είναι πολύ άριθμε φαντάζομαι και έτσι και εγώ προσπαθώ να βρω από πλευρά μου ένα συμβασμό αποδεκτό κυρίω ε, στο να ληφθούν υπόψη και οι ε, ανάγκε προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πολύ απλό ο λόγο για τον οποίο μείωσα από το 23% στο 20% και να σα εξηγήσω ότι δεν μπόρεσε κανεί μάλλον δεν, μπόρε, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσω συνένεση ως προς το ποιο θα πρέπει το σημείο εκκίνησης. Και άρα εγώ επέλεξα τη λύση της της μέγιστης δυνατή λύση που θα μπορούσα να δεχθώ για να δω στην συνέχεια και χάρη στη συζήτηση εάν αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα κοινό παρονομαστή για όλους. Και επίσης θέλω να επισημάνω ότι εδώ έχουμε πολλά προβλήματα να ξεπεράσουμε, πολλά εμπόδια και όχι μόνο νομικά νομικού χαρακτήρα, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε την πρώτη νομοθετική πρώτα στο πράσινο και τη δικασία της ε, συναπόφαση, της συνομοθέτηση μάλλον. Αλλά έχουμε και ζητήματα στα οποία θα πρέπει να έχουμε ισχυρά επιχειρήματα όταν έρθει η ώρα για τι ε, διαπραγματεύσει με την Επιτροπή και το Συμβούλιο και θέλω να έχω ένα περιθώριο κίνηση εκ μέρου τη επιτροπή. Θα δείτε επίσης την παρέκκληση για τα τέσσερα κράτη-μέλη με το ελάχιστο ποσοστό παραγωγής γάλακτος που θα επέτρεπε στις οργανώσεις παραγωγών να διαπρακάνουν συλλογικές διαπραγματεύσεις για ποσοστό μέχρι το 75% της παραγωγής και αυτό βέβαια αφορά τις μικρότερες χώρες που δεν μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά ή σημαντικά την ε, παραγωγή. Στη συνέχεια Έχουμε το 16 και το 20 για την ε, λειτουργία των συνεταιρισμών, όπου θεωρώ πως είναι σημαντικό να προστατευτούν οι αποδοτικές δομές όπου υπάρχουν και λειτουργούν σωστά στι ε, χώρες. Η Επιτροπή μας λέει ότι θα αποκλειστούν από το κείμενο όσο έχει αυτό τώρα. Παραμένει όμως κατά την άποψή μου, μια σύγχυση για το θέμα αυτό και γι' αυτό θα ήθελα να διευκρινιστεί η κατάσταση και ο τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί. Στο άρθρο 125 ε η διαφάνεια ε, απαιτεί μηνιαίες δηλώσεις. Αυτό για να έχουμε μια καλή ανάλυση της παραγωγής γάλακτος, τακτική ανάλυση παραγωγής γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ συμφωνώ και προσθέτω ότι θα πρέπει τα δεδομένα αυτά να αξιοποιούνται προς όφελος όλων των εμπλεκομένων φορέων και παραγόντων και θα πρέπει τα δεδομένα προσωπικού ή απόρριτου χαρακτήρα να γίνονται σεβαστά έτσι ώστε να ε, λειτουργεί ισόρροπα αυτή η ε, ωφέλεια από τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την προσφορά και τη ζήτηση. Στη συνέχεια δε, έχω κάνει κάποιες προτάσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν νομοθετικές επιπτώσεις επιδράσει, ε, αντίκτυπο, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να τι λάβει υπόψη η Επιτροπή. Μία έχει να κάνει με την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη στο των γαλακτοκομικών, με την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των ε, κονδυλίων όπου είναι διαθέσιμα και θεωρώ ότι θα πρέπει ο γαλακτοκομικό τομέα να εξετάσει με πολύ μεγάλη προσοχή και κυρίω με ορίζοντα την μέσο και μακροπρόθεσμη ε, βιωσιμότητα της, του κλάδου την αξιοποίηση των κονδυλίων. Και δεύτερον, έχουμε το σύστημα των υπείων ε, δανείων που θεωρώ ότι θα πρέπει να περιληφθεί μέσα στην έκθεση. και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθούν αυτά. αυτά. Δεν ξέρω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει τα κράτη εκείνα τα οποία αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες. Και επίσης δεν ήθελα να εξηγήσω τις τροπολογίες 9-11 και 21-40, στις οποίες έχουμε καταγράψει πιστεύω μια κοινή αντιμετώπιση στην οποία καταλήγουν τα θεσμικά όργανα εν ώψη της θέσης εφαρμογή του κανονισμού για τις ε, εφαρμοστικές πράξεις. Στην 179 τροπολογία 1 καταργώ το άρθρο, διότι διαγράφω μάλλον το άρθρο, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με εκτελεστικές πράξεις που αφορούν και τα καπνά, το οποροκυπευτικά και το καθεξής και εδώ θα πρέπει να έχουμε την λύση, ε, την εισαγωγή της λύσης με έναν οριζόντιο κανονισμό. Αντικαθιστώ το κείμενο με στην 172 με, την τροπολογία 22. Επίσης, διαγράφεται η παράγραφος 125 σχετική με τις συμβάσεις, 185 σχετική με τις συμβάσεις, στην ε, τροπολογία 23, διότι θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία της διαπραγμάτευσης, πρέπει να διαφυλαχθεί και να υπάρχει ένα λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστεί εγγυητή και να έχει δυνατότητα παρέμβαση σε αυτή την υπόθεση. Και επίση, κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι έχει ληφθεί ήδη απόφαση για ε, ε, να μπει ένα τέρμα στο σύστημα των ποσοστώσεων. Ίσως λοιπόν το ζήτημα της ήπιας προσγείωσης ή της ανώμαλης προσγείωσης ίσως να ε, πρέπει να το δούμε μέσα από αυτό το πρίσμα. Αυτό έχει να κάνει και με την κατεργασία των γαλακτοκομικών προϊόντων αλλά και με τους παραγωγούς. Και δεν πρέπει να λησμονήσουμε την λιανική, το τομέα της λιανικής, εκείνους δηλαδή οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν το κατά πόσον είναι ε, πικερδής η παραγωγή του γάλακτος. Και ξέρω τουλάχιστον από τη δική μου την παραγωγή και πείτε μου αν κάνω λάθος, ότι ο τομέας της λιανικής στο γάλα δεν, ε, τη ναι. χάνει τον ίδιο, δεν βρίσκεται ουσιαστικά υπό τον ίδιο έλεγχο με τον, το, τον οποίο υφίσταται ο τομέας της παραγωγής και της κατεργασίας. Και επίσης άλλη μία πτυχή ανησυχητική και την οποία μου εξέθεσαν ε, εκπρόσωποι που ήρθαν από την Ελβετία και που είχαν μεταπηδήσει από την ποσόστοση, και η οποία είχε μεταπηδήσει από την ποσόστοση στις συμβάσεις με σημαντική μείωση στην ε, παραγωγή και κατά 25% τουλάχιστον ε, μείωση του κέρδους του περιθωρίου κέρδους για τον παραγωγό. Χωρίς να θέλω να πω ότι θα επαναληφθούν ακριβώ τα ίδια. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφου ότι πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη να μην λησμονούμε τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε, με τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε την επιβίωση των ίδιων των μικρομεσαίων παραγωγών γαλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ευρώπη. Και κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι περιμένω να ακούσω τι απόψει των συναδέλφων στην ε, έκθεση αυτή και τι τροπολογίε του η προθεσμία που έχουμε είναι 22 Μαρτίου, δεν υπάρχει πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο. Πιστεύω όμως ότι έτσι θα μπορέσουμε εγκαίρως να επεξεργαστούμε συμβαστικές λύσεις πριν καταλήξουμε στην οριστική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από τον κύριο Νταντέν και κυρία Μπελακατούπρη. <coughs> Παρακαλώ, Μισελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα εξ ονόματος ομάδας μου να ευχαριστήσω τον Γιάννη Νίκολσον για όλη του την εργασία της συνεννοήσεις με τις άλλες ομάδες πριν συγγράψει την έκθεση του. Όλοι φαντάζομαι συμφωνούμε ότι το σύστημα έτσι όπως λειτουργήσε τελευταία δεν ήταν το καλύτερο δυνατόν. Αποφασίστηκε να καταργηθεί. Θα το αντικαταστήσουμε με ένα σύστημα συμβολέων και μας ανέφερε το παράδειγμα των Ελβετών ο Γιάννης. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε όλοι αυτό το παράδειγμα, αλλά στην ομάδα μου αναρωτιόμαστε μήπως δεν είναι δυνατόν με τα συμβόλαια και μόνο να γίνει καλή διαχείριση της αγοράς. Μήπως θα έπρεπε δηλαδή στην έκθεση αυτή να προβλέπετε και ένα ρήτρο αραντεβού για να κρίνουμε καλύτερα την αποτελεσματικότητα όσο μια ρήτρα αναθεώρηση να δούμε κατά πόσον δούλεψε καλά το σύστημα. Πρέπει ίσως να δώσουμε και στους παραγωγούς τη δυνατότητα, την προστασία να είναι σε θέση να διαπραγματεύονται πράγματι με τους πελάτες των και να μην ξαναβρεθούμε στην πραγματικότητα του 19ου αιώνα ή των αρχών του 20ου όπου ο παραγωγός είχε μπροστά του έναν αγοραστή παντοδύναμο. Ε, σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να ξεπεράσουμε λίγο αυτά που προτείνει η Κομισιόν και ο εισηγητής για τον καθορισμό, για τον ορισμό του ίδιου του συμβολέου και να δώσουμε περισσότερες εγγυήσεις στο διαπραγματευτή του συμβολέου ή τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να τύχει άνα διαπραγμάτευσης. Άλλο θέμα που τίθεται είναι η διαφάνεια έχουμε συνείδηση ότι πρέπει να υπάρξει εγγύηση της ασφαλείας των ε, νομικών πράξεων στο εμπόριο, αλλά για να μπορέσει κανείς να συνάψει ένα συμβόλαιο πρέπει να γνωρίζει καλά ποια είναι τα δεδομένα της συγκεκριμένη αγοράς και πρέπει να είμαστε νομίζω εδώ ανυποχώρητοι ως προς τις συνθήκες διαφάνειας και γνώσης των ενδιαφερομένων. Πράγματι η πρόταση της Κομισιόν αφορούσε ή ανέφερε το πρώτο δείγμα δηλαδή την σύναψη σχέσης μεταξύ γαλακτοπαραγωγού και αγοραστού ή αγοραστρίας. Αλλά ίσως πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό, τουλάχιστον ως προς τη διαφάνεια, γιατί είναι προφανές, ότι σε ολόκληρη την αγοραστική αλυσίδα επηρεάζονται τα έσοδα του παραγωγού και δυστυχώς το αφήνουμε και το λέω επίτηδες αφήνουμε όχι δίνουμε μόνο τα υπόλοιπα αυτό είναι απαράδεκτο και γι' αυτό πρέπει να είναι πιο αυστηρή όλη αυτή η διαδικασία πρέπει νομίζουμε η μέθοδος σύναψης αυτών των συμβολέων να είναι πιο ορατή από τον παραγωγό και τον αγοραστή, να σταθεροποιεί τα ε, έσοδα και να διέπεται από μια υγιή διαδικασία σύναψης συμβολέων. Άρα, σε όσα θα ζητήσουμε πρέπει να μιλήσουμε και για τα ποιοτικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Μας είχε πει το πρωί ο Επίτροπος ότι είναι ανοιχτός πριν λήξουν οι διαπραγματεύσεις αυτού των έννοια της ποιότητας. Το κείμενο μιλάει για διαχείριση των όγκων και των αγορών συμπεριλαμβανομένων μεταξύ των κριτηρίων και τα κριτήρια προέλευσης και ποιότητα και αυτό θα έπρεπε να το λέμε σαφέστερα στην εκθεσή μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μισόλ. Κύριε Σπέλη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι... προφανέ Σταραμπέλ, είναι προφανές ότι η έκθεση του κύριου Νίκολσον, του James, έρχεται σε ένα δύσκολο παγκοσμιοπλαίσιο, αλλά και σε ένα πλαίσιο που αλλάζει σε παγκοσμίο καθώς μέχρι σήμερα χάρη στις ε, ποσοστώσεις είχαμε σταθεροποιήσει τις ε, ποσότητες εξαγωγής ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν στραφεί προς την εσωτερική αγορά τώρα στρέφονται προς το εξωτερικό το λέω αυτό για να το έχουμε κατά νου στο μέλλον η αστάθεια αυξάθηκε και είδαμε ότι είχαμε στάθεια το 2008-2009 και θα επαναληφθεί και άλλες κρίσεις θα έρθουν στο μέλλον Μέχρι σήμερα σίγουρα εξαρτώνται οι τιμές παγκοσμίω από τη Νέα Ζηλανδία και την Οκεανία και από τις ποσότητες προς εξαγωγή. Και έτσι λοιπόν η κατάσταση απαιτεί τη, τη λήψη μέτρων, ισχυρών μέτρων ρύθμισης και να σας πω ότι εδώ και αυτή είναι η παρατηρήση επί της μας, δεν ε, βλέπω να υπάρχει βούληση για τέτοια ισχυρή ρύθμιση και νομίζω ότι το χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις καταρχήν να θέσουμε έμφαση, να δώσουμε έμφαση στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Ναι, σίγουρα είναι απαραίτητο, υπάρχει έλλειψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να αποκρύπτουμε την ουσία του προβλήματος ότι έχουμε την ε, ανισορροπία ε, σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής να αναφερθώ και σε κάτι το οποίο ανέφερε ο Τζέιμς. 33% έχουμε στην πρόταση. Ξέρω ότι υπάρχουν αποκλήσει. Στην πρόταση εγώ θα έλεγα να είμαστε πάνω από την Κομισιόν. Θα πρότεινα 80% και έτσι θα φτάναμε στο 50% κατά μέσο όρο. Δεν ξέρω τι θα πούν οι υπόλοιποι βέβαια. Εδώ μιλάμε για την ισορροπία μιας αγοράς, όμως ε, δεν υπάρχει ισορροπία στην ίδια την ε, έκθεση και καθώς έχουμε σχεδόν μονοπόλια, ε, έχουν ένα ισχυρό χαρτί διαπραγμάτευσης και για την τροπολογία 17 δεν κατανοώ τι εννοείται εδώ Δηλαδή, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία μεταξύ παραγωγού και μεταπητή. Αυτή η ισορροπία δεν υπάρχει. Θα πρέπει εμεί να την δημιουργήσουμε, να την αποκαταστήσουμε. Και γι' αυτό το λόγο Θέλω να πω ότι ο εισηγητής ε, προωθεί πάρα πολύ και παρουσιάζει ιδιαίτερα τη στρέβλωση του αγωνισμού. Κοιτάξτε, ε, ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε από τις αρχές να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και όχι να θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι το ιερό που δεν το αγγίζουμε. Δεν είναι δόγμα ο ανταγωνισμός. Ε, δεν ε, θέλω να μιλήσω εδώ τώρα για την αγορά ενέργειας, το έχουμε αναφέρει ήδη, όμως πολίτες ε, θα ήθελα να μην βλέπουμε τον ανταγωνισμό κάτω το ιερό. Θέλουμε να κερδίσει τελικά ο καταναλωτής για την τροπολογία 25, για μέγιστη ευελιξία. Ε, κοιτάξτε, δεν ξέρω. Ε, πρέπει να δούμε τι ακριβώς εννοούμε με αυτόν τον όρο ευελιξία. Όταν το ακούμε, τον όρο αυτό, εντάξει, μας ικανοποιεί πάντοτε, όπως και άλλοι όροι. Αλλά το θέμα είναι να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό στην πραγματικότητα. Και εδώ η ιδέα των συμβάσεων πρέπει να είναι ε, κάτι πάγιο, στέρεο. Πρέπει οι συμβάσεις να δίνουν μια ένδειξη του όγκου, των τιμών, ακόμη και ενδεικτικά, ακόμη και του τρόπου που καθορίζουμε τις τιμές και μιας διάρκειας ε, παραδείγματο χάρη, οι τιμέ ε, έχουν μια φόρμουλα. Θα μπορούσε να περιλαμβάνεται η εξέλιξη των τιμών, ε, των ε, τροφίμων ή του ζωικού κεφαλαίου. Γιατί εκεί έχουμε διαφοροποίηση στο κόστο παραγωγή. Διάρκεια. Επίσης σημαντικό μου φαίνεται να έχουμε μία διάρκεια ε, τουλάχιστον πρόθεσμα, γιατί διαφορετικά δεν ε, υπάρχει προβολή στο τομέα και δεν πρόθεσμα. συμβάσει δεν έχουν ε, νόημα. Όταν δανειζόμαστε την τράπεζα έχουμε ένα ποσό και ένα επιτόκιο για κάποιο διάστημα. Μπορεί να εξελιχθεί το επιτόκιο, το ίδιο και για την τιμή. Μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε μια ψαλίδα. Έτσι λοιπόν, εδώ θα πρέπει να συμμετέχει και η δημοσιαρχή και θα επανέλθω θα έλεγα λοιπόν ότι οι προτάσεις σε σχέση με τις συμβάσεις, ε, κοιτάξτε, θα ήθελα να είναι πιο ε, αυστηρά, όχι να έχουμε τόσο πολύ μεγάλη ευελιξία και να επανέρχεται, να αποκαθίσταται μια ισορροπία που έλειπε μέχρι τώρα. Τώρα στη διαπραγματευτική δύναμη αναρωτιέμαι αν ε, θέτουμε το ίδιο ερώτημα του σχεδόν μονοπωλίου για τους αγοραστές, όπως έχουμε στη Δανία στις κατοχώρες, ε, λόγου χάρη. Είναι σαφές, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε και στους παραγωγούς που είναι ο αδύναμος κρίκος σήμερα στην Ελισίδα να έχουμε μια πραγματική δύναμη στις διαπραγματεύσεις. Για τη διαφάνεια συμφωνώ με τον εισηγητή γιατί χρειάζεται πιο γρήγορη προσαρμογή στην αγορά. Αυτό είναι η τελευταία, το τελευταίο που μπορώ να προσάψω στις, στις ποσοστώσεις. Ίσως ε, λοιπόν πρέπει να δούμε το θέμα της προσαρμογής γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αν ε, δεν μιλάμε πλέον για ποσοστώσεις εντάξει, αλλά πρέπει πάντοτε να ελέγχουμε τον όγκο και να μην ε, εξαρτώμαστε από παρεμβάσεις δεν ε, μπορούμε πλέον να έχουμε τις τιμές που είχαμε το 80 για το γάλα και το βούτυρο. Και επίση θα ήθελα να αποδώσουμε ένα ρόλο στις δημόσιες αρχές. Ε, γιατί εδώ προωθούμε ε, το θέμα των αρχών, ίσως θα πρέπει να έχουμε μια δημόσια αρχή που να καθορίζει το περιθώριο και τις τιμές. Μιλάμε για το παρατηρητήριο των τιμών. Θα μπορούσε αυτό το παρατηρητήριο να πει δεν μπορεί η τιμή να πέσει κάτω από αυτό το ελάχιστο και ανάλογα με τις συνθήκες ε, φυσικά εξελίσσεται και η τιμή όπως ε, λέω παραπάνω. Έτσι λοιπόν ε, θα προτείνω ίσως και μια τροπολογία που θα επιτρέπει και στο κοινό είτε μέσω της Επιτροπής είτε μέσω των Υπουργείων των Κρατών Μελών να μπορεί να ασκεί και μια λειτουργία ρυθμιστική ελέγχου. Ορτ και κατόπιν Ähm, ευχαριστώ, Καταρχάς, ευχαριστώ τον κύριο Νίκολσον για την έκθεση, την οποία θεωρώ ευπρόσδεκτη, έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και αναφέρεται στο ζήτημα του να δοθεί μία επιλογή για τον παραγωγό να προμηθεύει σε παραπάνω από ένα γαλακτοκομείο τα προϊόντα του Πιστεύω ότι το να έχουμε μία βάση ισοδύναμη ή ίση αντιμετώπισης δεν είναι μια λύση εύκολη τη στιγμή που έχουμε πολύ διαφορετικές δομές στους ε, παραγωγούς και στις περιοχές. Εάν έχουμε φαρυπήρει ένα παραγωγό, ο οποίος σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή περιφέρεια έχει μονοπωλιακή θέση. Πώς μπορούμε να τον συμπεριλάβουμε σε μια βάση διαπραγμάτευσης. Θα ήταν κάτι το άδικο. Καλό θα ήταν λοιπόν να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τη δημιουργία μιας άλλης βάσης η οποία θα ανέτρεπε πάλι στις ισορροπίες της αγοράς. Δηλαδή θα, θα έκανε τελικά το αντίθετο προς το που επιδιώκουμε. Στο όσα είπε ο κύριος ε, Ταραμπέλα για τον προσδορισμό μιας ελάχιστης τιμής από μια αρχή. Ίσως θα πρέπει να αποφύγουμε μέτρα πολιτικής παρέμβασης στην αγορά τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι είναι αντιπαραγωγικά, ότι δεν φέρνουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Και γι' αυτό θα πρότεινα στις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις να προχωρήσουμε, όπως άλλωστε ορίζεται εν γέννη, και στην περίπτωση αυτή ε, με μια μελέτη στα πέντε χρόνια του πώς έχει λειτουργήσει το σύστημα. Άλλωστε έχει δεσμευτεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε αν αυτή η εντολή για, τη συνολική, ε, για τους συνολικούς χειρισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνεχιστεί ή όχι. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να δούμε ποια είναι η κατάσταση, να σχηματίσουμε άποψη και να διατηρήσουμε τον έλεγχο λίγο πολύ της κατάστασης ώστε να μην δώσουμε μια λευκό επιταγή και επαόριστον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό τουλάχιστον πρέπει να το πράξουμε. Επίσης, μετά την εκπνοή των ε, συμβάσεων, καλό θα είναι να έχουμε τη δυνατότητα της ευελιξίας για τον ε, προμηθευτή, όπως βλέπω εδώ ότι προβλέπετε, αλλά ταυτόχρονα και να προβλεφθεί η δυνατότητα για εθελοντική εκούσια ε, σύναψη συμβάσεως, όχι δηλαδή βάσει κάποιου προτύπου πρέπει ο καθένας να ακολουθήσει, αλλά να ε, μπορεί ο παραγωγός, εάν το επιθυμεί, να ε, έχει αυτή τη δυνατότητα σύναψη συμβάσεως και να τον ενισχύουμε, αλλά χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει κάποιο, κάποια σύμβαση, ε, κάποιο πρότυπο σύμβασης, αλλά να μπορεί να τη διαμορφώσει όπως θέλει. Εκεί δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που θα συνεχιστεί και στην υπόθεση αυτή. Θα καταθέσουμε και με τις δικέ μα τροπολογίες μας, αλλά πάντως ε, η κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο κύριο Νίκολσον είναι σωστή. Ευχαριστώ κύριε Ραιμερ. Σμιτ. Και μετά Χόισλινγκ. Εντάξει Χόισλινγκ. Κύριε Πρόεδρε, ε, μας δίνετε την εντύπωση ότι δεν με βλέπετε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, εκφράσω τώρα τη θέση ομάδα μου στην υπόθεση αυτή. Κυρίε και κύριοι, είναι ένα ε, υγρό τρόφιμο το γάλα ιδιαίτερη σημασία και βλέπουμε βέβαια και πόσο ζωντανά αναπτύσσεται αυτή η συζήτηση αυτή η συζήτηση η οποία έχει να κάνει ουσιαστικά με την απελευθέρωση των αγορών γάλακτος. Και ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή είναι, όπως λένε πολλοί ήδη, ότι ε, δεν υπάρχει κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα. Αυτό λένε πολλοί, αλλά για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, μπορεί μεν η τιμή να είναι κάπου στα 30 cents και άνω το λίτρο, αλλά περνάει η κρίση ο γαλακτοκομικό τομέα και είναι πολλοί οι παραγωγοί που αγωνίζονται για να επιβιώσουν. Δεν είναι τόσο ορόδινα τα πράγματα όπω κάποιοι θέλουν να τα λένε. Ευχαριστώ τον κύριο Νίκολσον για την έκθεσή του. Ευχαριστώ πολύ για την επιδίωξη για ανάπτυξη διαλόγου. Μας έδωσε και μια οπτική γωνία προς την Ελβετία για να μας υπενθυμίσεις ότι είναι πολλά αυτά που θα πρέπει να αποφεύγουμε να επαναλαμβάνουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Ίσως είναι συστήματα τα οποία δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο κύριος Νίκολσον, αλλά ίσως να μην πάνε τα πράγματα πάντα ε, όπως τα διαπιστώνουμε στην Ελβητία. Φερρυπίν μπορεί να μην ε, είναι καταστροφικές οι συνέπειες της κατάργησης των ε, ποσοστώσεων ίσως η Ευρώπη να έχει μια διαφορετική εξέλιξη. Δεν θέλω ωστόσο να υπογραμμίσω ότι είναι τόσο πολλά τα μονοπόλια στην Ευρώπη που ο παραγωγός δεν μπορεί καν να επιλέξει γαλακτοκομείο. Στη Γερμανία, στη Βόρεια Γερμανία παραδείγματι, είναι τέτοια μονοπωλιακή κατάσταση που δεν υπάρχει εναλλακτική. Δεν έχει ο παραγωγός επιλογή. Είναι μηδενικές οι εναλλακτικέ που προσφέρονται. Το ίδιο βλέπουμε και σε χώρες όπως η Δανία, που πάλι δεν υπάρχει δυνατότητα η εναλλακτική προσφορά. Άρα είναι πολύ περιορισμένο το περιθώριο χειρισμών ή κινήσεως του παραγωγού. Άρα καλό θα είναι να έχουμε ε, ως δεδομένη την αρχή ότι ο παραγωγός δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να ασκήσει πίεση στις διαπραγματεύσεις. Η επιλογή όμως του κυρίου Νίκολσον ως προς την συμμετοχή στις ε, συμβάσεις αυτές των παραγωγών δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει πόσο δεινή είναι η κατάσταση το 33, το 20, το 23% ε, των παραγωγών δεν είναι ποσοστό αποδεκτό για περιοχές όπου είναι πολύ υψηλή συγκέντρωση και η μονοπωλιακή θέση των γαλακτοκομείων, των γαλακτοκομικών παραγωγικών μονάδων. Και γι' αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ πιο μεγάλη προσοχή τον τρόπο με τον οποίο να αξιολογούμε τη διαπραγματευτική ισχύ του παραγωγού ή τη διαπραγματευτική ισχύ αντίστοιχα του συνεταιρισμού παραγωγών. Είναι λάθος επίσης να ε, εμπιστευτούμε για τα πάντα του συνεταιρισμούς, γιατί οι συνεταιρισμοί έχουν μερικές φορές ακολουθήσει επιλογές οι οποίες όχι μόνο δεν εξυπηρετούν το συμφέρον του παραγωγού, αλλά του αντίον ε, αποβαίνουν σ' όφελος των ε, μονοπωλίων και όχι των δικαιωμάτων του επιμέρους ε, μικρού παραγωγού. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις γαλακτοπαραγωγικές επιχειρήσεις. Η παρακολούθηση, η ιδέα για θέσπιση μιας υπηρεσίας επιτήρησης, monitoring, της κατάστασης της αγορές. Νομίζω ότι είναι χρήσιμη. Μπορεί μια τέτοια υπηρεσία να μας ε, καθοδηγήσει προς μια πιο ευέλικτη ε, προς ένα πιο ευέλικτο σύστημα χειρισμών της παραγωγής και της ζήτησης και μπορεί να είναι χρήσιμη εν τέλει. Και 7% λέτε ότι δεν ε, καλύπτεται ε, επαρκώς και ως εκ τούτου δεν είναι σωστός ο προσδορισμός ποσοστώσεων. Ε, ναι, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι είδους ε, προσφορά έχουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκής αγοράς. Δεν έχει κανένα νόημα λοιπόν η ποσόστοση όταν έχει τόσο χαμηλή απορρόφηση. Και επίσης δεν ρεσμονούμε ότι πριν το 2014 θα κληθούμε για άλλη μια φορά να ασχοληθούμε με το θέμα του γάλακτος, αλλά αν περιμένουμε μέχρι τότε θα είναι πολύ αργά να ε, εξετάσουμε εκ βάθρων το σύστημα. Δεν πρέπει να περιμένουμε το 2014-2015. Πρέπει πολύ νωρίτερα να μελετήσουμε το τι θα πράξουμε όταν καταργηθούν οι ποσοστώσεις. Ποιε θα είναι οι συνέπειες για, την, ε, όλη, για τον όλο κλάδο. Δεν θα είναι πιστεύω τόσο εύκολα τα πράγματα και θα έχουμε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ Μάρτιν, ο κύριος Χάσπορτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκολσον για την έκθεσή του και να τον υποστηρίξω. Όμως πιστεύω ότι υπάρχουν ε, δύο προβλήματα στον τομέα στο οποίο θέλω να αναφερθώ καταρχήν ένα πρόβλημα που χρησιμοποιείται από την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον τομέα του γάλακτος. Το γάλα έχει ένα ιστορικό ότι είναι σε υπερπροσφορά, είναι μια πρωτήλη και παρά το ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κατακαιρματισμός ε, μεταξύ προϊόντων ε, υψηλής αξίας και χαμηλής αξίας. ή. Ε, ε, τιμή που πληρώνεται ε, στους ε, παραγωγούς πάντοτε θα φέρει την τιμή ενός προϊόντος ακατέργαστου πρώτης ύλης. Η παραγωγοί δεν έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν την προσφορά και τη ζήτηση, ούτε την τιμή που λαμβάνουν και ε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τελικά να μην καθορίζουν οι ίδιοι τις τιμές, αλλά να δέχονται αυτό που τους δίνουν ως τιμή. Δεύτερον, ε, έχουμε και κάποια προβλήματα από την πλευρά της προσφοράς, ε, γιατί ε, καταρχήν οι παραγωγοί αρνούνται στον εαυτό τους να προσθέσουν αξία στην παραγωγή τους και έτσι λοιπόν εκτίθενται ακόμη περισσότερο στις ανισορροπίες στην διατροφική αλυσίδα, αλλά όπως και οποιοδήποτε άλλο ε, αγαθό πρώτης ύλης, ε, η απάντηση των παραγωγών στις χαμηλές τιμές είναι να αυξήσουν την παραγωγή. Αυτό το κάνουν γιατί δεν δημιουργούν ανεναλλακτική για τον εαυτό τους και έτσι λοιπόν απλώς αυξάνουν την παραγωγή και φυσικά αυτό ξύνει το, πρόβλημα που προσπαθούν να αποφύγουν. Έτσι λοιπόν, ε, ενώ καλωσορίζω τις προτάσεις του κ. Νικολσόν, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ρεαλιστέ για το τι μπορούμε να πετύχουμε. Και θέλω να τονίσω ότι αυτέ οι δράσει μπορούν να βοηθήσουν τον τομέα μόνο αν ο τομέας είναι σε θέση και είναι έτοιμο να βοηθήσει τον εαυτό του. Με εκπλήσει το ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ή αδικίες στον τρόπο που λειτουργούσαν οι συμβάσει στον τομέα του γάλακτο είναι από την πλευρά τη ε, προσφορά. Υπάρχουν πάρα πολλέ υποχρεώσει χωρί να υπάρχουν εγγύησει για την τιμή που πληρώνεται ενώ το μέσο τη μεταποίηση έχει την ικανότητα να αλλάξει την τιμή κατά τη δική του διακριτική ευχαίρεια, χωρί ε, καμία αναφορά ε, στην ε, πλευρά τη προσφορά. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν οποιοδήποτε αλλαγέ στι τιμέ που περνούν κατευθείαν στον παραγωγό και ο παραγωγό πρέπει να απορροφήσει όλο τον κίνδυνο του τομέα, ενώ πολύ λιγότερο απορροφά η πλευρά του αγοραστή. Έτσι λοιπόν υποστηρίζω τι προτάσει του James για τι συμβάσει, υποστηρίζω τη ρήτρα αποκλειστικότητε, αλλά και πάλι πιστεύω ότι οι εναλλακτικέ ε, είναι. Ε, πολύ ε, λίγες και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις συμβάσεις. Επίσης αναγνωρίζω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ανταγωνιστικότητα στον ε, γαλακτοκομικό τομέα και οι αναγκαστικές συμβάσεις μπορεί να χρειάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά εδώ θέλω να τονίσω ότι αυτή την απόφαση πρέπει να την πάρουν τα κράτη-μέλη. Είναι ένα θέμα επικουρικότητας. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκολσον για την εκθεσή του και να εκφράσω την υποστήριξή μου. Για να συνεχίσουμε τώρα, κύριος Άλμπερτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω από την αρχή της σου, Γνωρίζω όμως αρκετά καλά την έκθεση του κυρίου Νίκολσον. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που ανέλαβε αυτό το δύσκολο έργο. Γνωρίζω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να δώσει εδώ λύσεις στα θέματα αυτά. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και πανάκιες και γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να βρούμε μια λύση. Δεν θα είναι εύκολο. Θα ήθελα να δώσω κάποιες ε, ενδείξεις στον κύριο Νίκολσον για τα πράγματα που με ενδιαφέρουν. Έχουμε Έχω συμμετοχή σε μια γαλακτοκομική μονάδα η οποία λαμβάνει γάλα από 7.000 διαφορετικούς βαβαρούς ε, παραγωγούς γάλακτος. Ε, έχουμε λοιπόν το εξής πρόβλημα, ότι δεν είναι χαμηλές ε, οι τιμές του γάλακτος, υπάρχει, υπάρχει βέβαια δυνατότητα μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα παραγωγού των προμηθειών σε γάλα, υπάρχει περιπθώριο για περισσότερες πιέσεις και, είμαστε, και είναι υποχρεωμένος παραγωγός να πουλήσει. Γι' αυτό λοιπόν θα σκοπίμω να προσδοριστεί ένα χρονικό όριο το οποίο να ορίζει την, ε, τον επαναπροσδορισμό της τιμής ε, το πολύ μέσα σε έξι μήνες. Να μην Ξεπερνά δηλαδή το διάστημα για το οποίο ισχύει αυτή η σύμβαση το εξάμεινο, διότι διαφορετικά, εάν είναι η τιμή χαμηλή, μπορούμε να έχουμε ε, μια σύμβαση ενό έτου φερρυπίνη. Εάν όμω είναι αρκετά υψηλή η τιμή, τότε δεν θα δέχεται ο παραγωγό άλλη σύμβαση από τετράμινη και χαμηλότερη. Και γι' αυτό δεν μπορεί να δουλέψει αποτελεσματικά μια γαλακτοπαραγωγική μονάδα. Μπορούμε να πούμε, αφού θα υπολογίζουμε θα αρχίσει να εφαρμόζεται από Σεπτέμβριο η, ε, μια τέτοια σύμβαση, ότι θα ισχύει μέχρι τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους και ότι έτσι θα μπορεί κανείς να υπολογίσει ε, τις προμήθειές του χωρίς ε, πολλές πιέσεις. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε λοιπόν τουλάχιστον ένα εξάμεινο διάρκειας αυτής της σύμβασης. Και χωρίς αυτή την ε, προθεσμία, εάν δεν την ορίσουμε, δεν θα μπορεί ο κλάδος της κατεργασίας του γάλακτος, ακόμη και με ένα εκατομμύριο τόνους ε, ε, γάλακτος, να επηρεάσει, να διεκδικήσει αυτά τα οποία θα ήθελε σε μια σύμβαση με τους παραγωγούς. Επίσης, το ίδιο θα έπρεπε να ορίσουμε ε, προθεσμίες για την καταβολή των στόχων πληρωμής από τη λιανική, από τις αλυσίδες δηλαδή ε, μεταπόλησης, 40, 60, 80 μέρες, που θα επιτρέπουν την ενδιάμεση χρηματοδότηση των γαλακτοπαραγωγικών μονάδων. Διότι διανοηθείτε, όταν έχουμε γάλα φρέσκο, ημέρα που λέμε, το οποίο έχει πολύ μικρή διάρκεια ζωής, ε, πρέπει να κατανοηθεί μέσα πολύ λίγες μέρες, ε, το να ορίζεται σε μια σύμβαση ε, μεταπόλησης ότι η αμοιβή θα δοθεί 60, 70, 80 μέρες αργότερα είναι καταστροφικό διότι θα πρέπει ε, ή να δεχθεί κανείς μια τέτοια λύση είτε να αρνηθεί και τότε το προϊόν του το έχει χάσει. Δεν έχει περιθώριο δηλαδή να διαπραγματευτεί με κάποιον άλλον την πόλη του προϊόντος. Και δεν είναι νοητό βέβαια να παίρνουμε την, ε, το τίμημα ενός προϊόντος το οποίο έχουμε πωλήσει σήμερα μέσα σε δύο-τρεις μήνες ή περισσότερο. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, να περάσω και στο θέμα των συνεταιρισμών, γιατί απαιτούμε αφενός οι οργανώσεις, η ε, παραγωγή ε, να οργανώνονται. Εάν όμως οργανώνονται σε πολύ μεγάλο συνεταιρισμό, ε, τότε αντιδρούμε γιατί λέμε αυτό είναι μονοπόλιο του συνεταιρισμού και δεν είναι καλό πράγμα και δεν το θέλουμε. Ε, ναι, αλλά κοιτάξτε να σας πω, εάν πρόκειται για ένα συνεταιρισμό γεωργών και συμμετέχουν όλοι οι γεωργοί, όλοι οι παραγωγοί σε αυτό το συνεταιρισμό, πρόκειται για ένα συνεταιρισμό που 100% ανήκει στους παραγωγούς. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί συμμετέχουν με τα, μέσα στα όργανα τα, τα διοικητικά και λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις είναι καθαρά οργανώσεις παραγωγών αυτοί οι συνεταιρισμοί. Ναι, ναι, ναι. Εάν δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, αυτό οφείλεται μόνο γιατί, γιατί κάποια επιμέρους μέλη του ενδεχομένω έχουν ισχυρότερη θέση και επηρεάζουν τα πράγματα. Οπότε είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ορισμού ο συνεταιρισμό θα πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε όπως ακριβώς και τον κάθε παραγωγό. Ευχαριστώ πολύ. cuvântul Κυρία Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Νίκολσον για την εργασία του. Από τη δική μου οπτική Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για δράση. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι εξακολουθεί να αξίζει τον κόπο να επιμείνουμε επί ορισμένων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ε, όπως σας είπα, πραγματικά προκαλεί σύγχυση και Πραγματικά δεν θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, δεν θα δώσει κατάλληλη απάντηση στα προβλήματα που έχει ο τομέας για την προοπτική του τέλους των ποσοστώσεων για το 2015 και να ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Η έκθεση παρουσιάζει το τέλος των ποσοστώσεων ε, ως κάτι δεδομένο και δεν φαίνεται να είναι λογικό κάτι τέτοιο δεν ε, το θεωρώ λογικό γιατί τελικά έχουμε μία πρόταση της ε, Επιτροπής ως εναλλακτική αλλά πρέπει να δούμε καταρχήν αν λειτουργεί αυτή η πρόταση ως εναλλακτική. Αυτό που έχουμε ενώπιόν μας ε, δεν οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ΕΚΟΜΗ και η ίδια Επιτροπή φαίνεται ότι το αψηφά αυτό γιατί προβλέπει μία εκτίμηση, μία ε, αναθεώρηση του ίδιου του συστήματος των συμβάσεων για το 2014. Έτσι λοιπόν χρειάζεται και εμείς να μπορούμε να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα των προτάσεων αυτών που έχουμε τώρα επιτάπητος, να δούμε πώς λειτουργήσει επιτόπου και το 2014 έχουμε ανοιχτεί την πόρτα έτσι μέσω της αξιολόγησης να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ρύθμισης στο τομέα. Ναι. Κατόπιν πιστεύω ότι εδώ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σόφρονες ε, και να μην ακολουθούμε την ε, προσέγγιση όπως ε, η προσέγγιση που βλέπουμε στις τροπολογίες 3, 6, 12 και 28. Θα έπρεπε να είμαστε πιο σόφρονες γιατί ουσιαστικά εδώ ανοίγουμε την πόρτα για αυτή την δυνατότητα αναθεώρησης που προτείνει και η Κομισιόν για το 2014. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μας παρουσιάζει το εξή. Αφήνει εκτός το θέμα της διανομής και εμείς όλοι έχουμε την εντύπωση ότι αν αφήσουμε εκτός τη διανομή πάντοτε η πρόταση αυτή θα είναι ακροτηριασμένη, θα είναι κουτσή και αυτό είναι ακόμα λόγος που αιτιολογεί την λίγη πίστη που έχω εγώ στην πρόταση αυτή. Δεν πιστεύω ότι θα επιλύσει τα προβλήματα του τομέα, δεν πιστεύω ότι θα εγγυηθεί μία βιώσιμη ανάπτυξη για τον τομέα σε όλα τα κράτη-μέλη όπου αυτή τη στιγμή τίθεται σε εφαρμογή. Αν αφήσουμε τη διανομή εκτός δεν έχουμε ιδιαίτερε λύσεις εδώ. Ε, εγώ νομίζω ότι σε αυτή την έκθεση πρέπει να τονίζουμε την αναγκαιότητα να συμμετέχει εδώ και ο τομέας της διανομής. Δεν μπορούμε να δεκτούμε τη θέση του Επιτρόπου που λέει ότι ε, δεν εντάσσεται εδώ η διανομή. Πρέπει να είμαστε δημιουργική, να βρούμε τρόπους, ε, να ασκήσουμε πίεση έτσι ώστε και η διανομή να μπορεί να ε, συμμετέχει όταν θα σταθμίζουμε τις λύσεις για τον τομέα, ακόμη και στις διακλαδικές οργανώσεις. Δηλαδή, εδώ να αναφέρουμε μοντέλα για τις διακλαδικές οργανώσεις που να ε, λειτουργούν ε, όπως ε, είναι το συμβουλευτικό όργανο για το τομέα του γάλακτος και να συμμετέχει όλος ο τομέας. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι παρούσα και διανομή εδώ. Διαφορετικά δεν θα καταλήξουμε πουθενά με αυτές τις προτάσεις. Επίσης, νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε στη δημιουργία του παρατηρίου για τον καθορισμό των τιμών, γιατί όλοι θεωρούμε ότι η τιμή στον παραγωγό ε, δεν ανεβαίνει, όταν ανεβαίνει δεν ανεβαίνει επαρκώς, δεν αυξάνεται επαρκώς η τιμή σε σχέση με αυτό που δεν βλέπουμε να συμβαίνει κατά μήκος της αλυσίδα και βλέπουμε κάποια στιγμή να αυξάνονται τα σιτηρά τόσο πολύ και πάνω από τα καύσιμα παραδείγματος χάρη. Έτσι λοιπόν ε, δεν υπάρχει καμία αντιστάθμιση, κανένα ε, εισόδημα στον παραγωγό. Έτσι λοιπόν είναι λανθασμένο λέμε ότι είναι σταθεροποιημένο ο τομέα Αντίθετο, αυτό που βλέπουμε είναι ότι κλείνουν όλα και περισσότερες εκμεταλλεύσεις ε, και εγκαταλείπουν η παραγωγή τη δραστηριότητα αυτή. Θα ήθελα ακόμη να στήσω την προσοχή σας ε, σε αυτήν την υποτιθέμενη λύση με τις συμβάσεις. Ε, θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η πρόταση που μας υποβάλλεται ίσως ε, να είναι καλή για ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά δεν μπορεί να προσαρμοστεί στι ανάγκε όλων των κρατών μελών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση και το καθήκον να παρουσιάσει λύσει που να είναι λύσει ευέλικτε για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για διαφοροποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, να επικεντρωνόμαστε σε ορισμένα κράτη-μέλη και σε ορισμένου τομεί. Αυτό δεν έχει νόημα. Όταν βλέπω εδώ σε αυτή την πρόταση κυρίω συμβάσει. τι συμβάσει εκούσιε. δηλαδή όλα τελικά δεν καταλήγουν πουθενά. Γιατί ε, τα, κάποια κράτη-μέλη έκαναν συμβάσει, κάποια άλλη όχι. Γιατί αλλάζει λοιπόν. Αρχίζουμε να συζητάμε το θέμα του όγκου της διάρκειας. Γιατί γνωρίζουμε ότι σε ό,τι αφορά τη διάρκεια ε, είναι αυτό που είπε ήδη ο συνάδελφος. Δηλαδή δεν ε, κατορθώσαμε να πετύχουμε τη συνένεση μεταξύ των παραγωγών και των βιομηχανιών μεγάλες προθεσμίες για τις συμβάσεις. Ε, δηλαδή αυτό σε τι εξυπηρετεί αν είναι πολύ μεγάλη η αστάθεια των δημών και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι στην περίπτωση της Πορτογαλίας εμείς Κοιτάξτε, θα, κλείσω, θα κλείσω σε λίγο. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, το 70% δεν υπολόγισα σωστά το χώρο, με συγχωρείτε, θα το πω γρήγορα. Το 70% του πορτογαλικού γάλακτος ε, το παραδίδει η ίδια βιομηχανία. Δηλαδή, ε, σχεδόν μιλάμε για ένα μονοπόλιο, έτσι λειτουργούν οι συμβάσεις. Και για να κλείσω, μιλήσατε και για soft landing. Δεν νομίζω ότι θα είναι δυνατή αυτή η ομαλή προσγείωση, αλλά τουλάχιστον πρέπει να έχουμε πιο ε, μικρές συνέπειες. Πρέπει να προβλέψουμε ε, μία αποζημίωση για ορισμένους παραγωγούς ε, και πρέπει να προβλέψουμε συγκεκριμένα μέτρα για τις πιο ευάλωτες περιοχές, τις λιγότερο ευνομένες περιοχές που αποκλειστικά εξαρτώνται από την γαλακτοκομική παραγωγή. Με συγχωρείτε, μου ξέφυγε ο χρόνος, αλλά πρέπει να παρέμβω για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σερμπαρές. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νίκολσον για το έργο του και είναι πάρα πολύ δύσκολο το αναγνωρίζουμε. Ο κανονισμό, αναφέρεται στις συμβατικές σχέσεις ε, για το γάλα και για τα γαλακτοκομικά. Όμω η αλήθεια είναι ότι ε, στη συνέχεια αναφέρεται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των παραγωγών ε, ε, και ε, του, της βιομηχανίας δηλαδή ε, υπάρχει ουσιαστικά εδώ ένας ακροτηριασμός γιατί δεν καλύπτονται οι όλοι. Εμείς τα τελευταία 8 χρόνια εργαστήκαμε σε ένα συνεταιρισμό, ε, διαχειριζόμασταν ένα συνεταιρισμό μεταποίησης, ε, πρόκειται για ένα μεγάλο συνεταιρισμό που κάλυπτε 11 άλλους συνεταιρισμούς και ε, ουσιαστικά ε, πληρώναμε τα χρήματα και εκεί διαπραγματευόμαστε και συμβάσεις και με τη διανομή από τον Ιούνιο στο Δεκέμβριο είδαμε αύξηση ε, στις τιμές ε, πάνω από 39%. Ε, το γάλα αυξήθηκε 4,7 και το κρέας 3,6 και τότε αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι για να έχουμε μία ανάλυση των μέτρων που χρειάζεται το μέσο του γάλακτος έπρεπε να ξεκινήσουμε από την παραγωγή οποίο ε, πήγαμε ε, στα σημερινά σούπερ μάρκετ και αν πάμε στο σούπερ μάρκετ και δούμε πόσο πληρώνουμε το γάλα σήμερα είδαμε ότι βρισκόμαστε βρισκόμαστε ενώπιον ε, ενός προβλήματος που είναι το εξής. Ε, έχουμε τεράστια αύξηση της παραγωγής, ε, αλλά είναι διαφορετική, πολύ πιο υψηλή τιμή του γάλακτος στην κατανάλωση. Δηλαδή, όταν συνάπτουμε τις συμβάσεις, κατανοούμε ότι εδώ ε, διακυβεύεται και το θέμα της ε, σωστής ε, διανομής. Έτσι λοιπόν τιμή, διανομή και εισόδημα είναι θεμελιώδη. τώρα, εδώ... μιλάμε για τις συμβάσεις, Έχουμε επίσης μια καλή συνεισφορά για την παραγωγή και για το διακλαδικό τομέα, αλλά πρέπει να μπορέσουμε να καθορίσουμε αυτή τη ρύθμιση, δηλαδή να μπορέσουμε να δώσουμε ορθές τιμές και να εγγυθούμε και τους όγκους για το μέλλον. Δεν ε, αναφέρεται εδώ με σαφήνεια τι θα συμβεί αφού απορριθμίσουμε την αγορά με τις ποσοστώσεις και δεν ε, αναφέρεται ε, ποιες προοπτικές θα έχουμε για το μέλλον χωρίς αυτό το καθεστώς. Και αν είναι βέβαιο ότι οι συμβάσεις θα μπορούν να επιτρέψουν σε ορισμένους να δυσφαλίσουν κάποιες τιμές, δεν θα επιτρέψουν μέσα φήνεια την παραγωγή σε διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτό όμω είναι, πρέπει να το καλύψουμε, όχι ίσως αυτή την έκθεση, αλλά πρέπει να θέσουμε αυτό το πρόβλημα και πρέπει να το θέσουμε σε αυτή τη βάση. Ο τομέας αρχίζει στην παραγωγή και τελειώνει στην αγορά. Δηλαδή ε, πρέπει να έχουμε μια καθολική προσέγγιση και να δούμε τις θετικές πτυχές. Σας ευχαριστώ continuare are cuvântul domnul δέχομαι και εγώ αυτή την έκθεση και συγχαίρω τον κύριο Νίκολσον για όλα όσα έκανε καθώς και για την καλή του θέληση και συνεννόηση με όλες τις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν. Ως προς τα συμβόλαια και το πούλινγκ του γάλακτος. Συμφωνούμε απόλυτα και εμείς στη χώρα μου ότι το συνεργατικό κίνημα στην Ιρλανδία, γιατί το συνεργατικό κίνημα στην Ιρλανδία είναι ιδιαίτερα σημαντικό και συμβάλλει στη σταθεροποίηση της αγοράς. Δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά στην εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό, αλλά πάντως η διαφάνεια στις αγορές είναι κάτι ουσιώδες. Νομίζω ότι η πραγματική δυσκολία και το αδέχεται και η ίδια η Κομισιόν είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς τι θα κάνει η αγορά. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, αν μπορούσε να γίνει και εφαρμοζόταν θα ήταν θετικό φυσικά. Επίσης όμως πρέπει να δούμε, να πάρουμε μαθήματα από την εμπειρία του 2009 Βραχυπρόθεσμα καλά δείχνει να λειτουργεί η αγορά, αλλά δεν έχουμε καμιά εγγύηση γι' αυτό ότι δεν θα επαναληφθεί η κρίση του 9. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν υπήρχε, τι θα είχε γίνει αν είχε υπάρξει κάποιο δίκτυο ασφαλείας τότε το 9. Αν δεν υπήρχε δε κανένα όριο στην παραγωγή, επίσης φανταστείτε τι θα είχε γίνει. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε προβλέψει σχεδόν τίποτα για να αποφύγουμε την επανάληψη μιας τέτοιας κρίσης. Από την εμπειρία της χώρας μου θα έλεγα ότι υπάρχει βία, σημειώνεται μια βία να επεκταθεί, να αυξηθεί ξανά η παραγωγή. Ξέρω ότι η έκθεσή σας δεν αναφέρει αυτά τα θέματα, αλλά αυτή η βία για για αύξηση της παραγωγής, ε, αν δούμε ποιο είναι κόστος αντιπροσωπεύει, μπορεί να δημιουργήσει φόβους για κάποιον υπερφόρο που να καταλήξει μέχρι και στα 28,5 λεπτά το λίτρο. Στη χώρα μου έχουν ήδη αρχίσει να μιλάνε για τέτοιου είδους αυξήσεις. περίπου 7 με 8% των Ευρωπαίων παραγωγών εξαρτώνται από την ποσόστοση και είναι προφανές ότι οι τιμές των Δημητριακών, το κόστος ενοικίασης της γης και οι διεθνείς αλλαγές Μπορεί να μην μας επηρεάζουν άμεσα, αλλά έμεσα μας επηρεάζουν. Η παραγωγή ενός λίτρου γάλακτος σήμερα είναι 4 λεπτά ακριβότερη από ό,τι πριν από 3 χρόνια, α, χρόνια. Κοστίζει 8 λεπτά και η στήριξη φτάνει τα 20. Τι μέτρα λοιπόν μπορούμε να φανταστούμε στο μέλλον. Αν φυσικά στηρίξουμε έναν παραγωγό θα χρειαστεί να στηρίξουμε και τον χείτονά του, ο οποίος αν δεν έχει άλλη στήριξη θα γυρίσει και αυτό στην ίδια παραγωγή. Η έκθεση νομίζω είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα έπρεπε η Κομισιόν να δει και μεταξύ του 11, όχι μόνο το 11 με 15 αλλά και περαιτέρω τι θα γίνει. Διότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ε, διανομέων, των αγοραστών του γάλακτος δηλαδή. Ευχαριστώ. Πώς, πώς. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τις παρεμφάσεις. Έγινε συζήτηση. Ίσως η Επιτροπή θέλει κάτι να προσθέσει. Παρακαλώ. Κύριε Σπίσα Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι, ε, πολύ στόμος για να μπορέσουν να μιλήσουν και άλλοι συναδελφοί. Συγχαίρω τον ε, James Νίκολσον, που βλέπω έχει χρησιμοποιήσει ακόμη και το, το επίσημο όνομά του για την έκθεση. Ε, έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε όχι μόνο με την εικόνα αλλά και με τις δομές και υποδομές του τομέα του παραγωγής γάλακτος. Πολλά είναι τα προβλήματα που πρέπει να περιγράψουμε και να αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτό που με απασχολεί εμένα καθώς είμαι δικηγόρος κυρίως είναι η νομική ε, διάρθρωση του τομέα των γαλακτοκομικών η οποία είναι αποτρόπαια θα έλεγα και χωρίς νομική βάση δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τίποτα. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να δοθεί έμφαση σε αυτό. Θα ήθελα να είναι υποχρεωτικέ οι συμβάσει για όλα τα κράτη-μέλη δυνατόν και επίσης δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να αποκλείονται οι συνεταιρισμοί από την υποχρέωση για ε, σύναψη εκκίνηση διαπραγματεύσεων και σύμβαση, σύναψη συμβάσεων. Όλα αυτά στη τελευταία ανάλυση θα καταστήσουν ακόμη πιο διαφανή, ε, μετρήσιμη και απρόσκοπτη τη λειτουργία της ιστορικής αγοράς. Δεν έχει κανείς λόγο να φοβάται τις συμβάσεις, ε, αρκεί να είναι υποχρεωτικές για τους συναδέλφους που ζητούν πιο αξιόπιστα στοιχεία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στις ε, διαπραγματεύσεις του τελευταίου προπολογισμού είχαμε μιλήσει για την ανάγκη για ένα παρατηρητήριο τιμών που ήδη υπάρχει τώρα και μπορεί να μην είναι, είναι σε πιλωτικό στάδιο, μπορεί να μην είναι ε, πολύ δημοφιλές, αλλά πάντως βοηθάει και στον προγραμματισμό και στην αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων. Κατά τα άλλα, ε, ε, υποστηρίζω και εγώ τον κύριο Νίκολσον για την, στην έκθεσή του. Ευχαριστώ, Κουτιέρης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομο. Η κυρία Πετρέων είπε ότι ίσως αυτή η πρόταση, αυτή η έκταση να μην αρκεί. Και μάλλον έχει δίκιο στο ότι τίποτα δεν αρκεί, αλλά είναι όλα απαραίτητα για να βελτιώσουμε τις συνθήκες ε, και την διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών στη διατροφική λυσίδα. Εγώ θα ήθελα να κάνω ορισμένα επιμέρους σχόλια για την έκθεση Νίκολσον, καταρχήν. Να αναφέρω μια προσωπική ανησυχία σχετικά με το άρθρο 127α παράγραφος 5. Στο άρθρο αυτό εισαγάγεται μία εξαίρεση στις ε, αρμόδιες εθνικές αρχές για να περιορίσουν τη διαπραγματευτική ισχύ των οργανώσεων των παραγωγών για να αποφευχθεί ο αποκλεισμό, ε, όπως ε, λέει η Κομισιόν, ή σοβαρή στρέβλωση στον ανταγωνισμό, όπως λέει η τροπολογία του κυρίου Νίκολσον. Κοιτάξτε, ούτε το ένα κείμενο μου κάνει, ούτε το άλλο. Ούτε της Κομισιόν, ούτε του κυρίου Νίκολσον. Γιατί νομίζω ότι είναι σοβαρό λάθος να αφήνουμε τόσο μεγάλο περιθώριο ερμηνείας ε, στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνουν οι εθνικές αρχές είναι ερμηνεύουν και όλοι γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια ερμηνείας αναχώρα και νομίζω ότι έτσι προκαλούνται πολύ σημαντικές αποκλήσεις στο εμπόριο και σημαντικές ανισότητες στις ευκαιρίες που έχει ο ένας παραγωγός ή ο άλλος, ανάλογα με το πώς γίνεται ερμηνεία από τις αρχές ανταγωνισμού στο κάθε κράτος μέλος. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι το καλύτερο είναι να διαγράψουμε την παράγραφο αυτή ή να αναφέρουμε ποια όρια μπορούν να υπάρξουν ε, στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Ε, τώρα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη που επιλέγουν την υποχρεώθηση τικό χαρακτήρα των συμβάσεων να ε, αποκλείσουν ε, τις ε, μεταφορές όπου δεν συμμετέχουν οι παραγωγείς. Γιατί αν δεν το πράξαμε αυτό θα είχα, ε, αν το πράξουμε αυτό θα έχουμε πολύ μεγάλο ε, γραφειοκρατικό άχθος που δεν θα μπορούσε να σηκώσουν πολλά κράτη-μέλη και δεν θα υπήρχε καμία προσθέμενη αξία για την ενίσχυση των παραγωγών. Και σε μια συζήτηση όπου πάντοτε λέμε πόσο σημαντική είναι η απλούστευση της ΚΑΠ ε, και της γραφειοκρατίας, νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα μας βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων. Και ε, ο κύριος Τερεβέλα αναφέρθηκε στην τροπολογία 17 δεν ε, έγινε κατανοητό γιατί το 33% κατεβαίνει στο 20% σε αυτή την τροπολογία. Εγώ νομίζω ότι μπορεί εδώ ε, να μην ε, μπορέσουμε τελικά να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών. Εγώ νομίζω το 33% ήταν ένα νούμερο στο οποίο κατέληξε το Συμβούλιο συνενετικά. Ε, και κατόπιν συμβιβασμού. Έτσι λοιπόν αν αλλάξει κάτι τέτοιο χωρίς να το αιτιολογήσουμε ορθώς θα μπορούσε να παρουσιάσει πάρα πολλά προβλήματα. Και τέλος, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε τον ορισμό της ε, οργάνωσης παραγωγών ε, στο κείμενο που προτείνει η Επιτροπή ο ορισμός που μας παρουσιάζεται είναι πολύ γενικός, έτσι λοιπόν θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε έναν ορισμό παρόμοιο με αυτό που έχουμε στο 126 της ενοποιημένης εκδοχής ε, της ΚΟΑ που λέει πολύ σύντομα ότι οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να είναι αυτές που αποτελούνται από παραγωγούς ε, που δημιουργούνται με δική τους πρωτοβουλίου και που επιδιώκουν συγκεκριμένους στόχους και αναφέρονται κάποιοι στόχοι στον ίδιο τον κανονισμό. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλό να αγαγουμε αυτό σε αυτό το κείμενο για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Σας ευχαριστώ. Στεφάν Λεφόλ. Θα πράξω όπως μπορεί. Θα αναγγείλω ότι θα είμαι σύντομο, αλλά δεν ξέρω θα τα καταφέρω. Πάντω θέλω να ευχαριστώ τον Τζέιμ. Έκανε, ανέλαβε μεγάλο έργο. Τον ε, συγχαίρουμε. Αλλά πάντα σε τέτοιου συζητήσει υπάρχει η δυσκολία του να διαλέξουμε ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε περισσότερο την ανταγωνιστικότητα ή να καταπολεμήσουμε από την άλλη την πτυτικότητα των τιμών. Τον παραγωγό δηλαδή ή τον κλάδο της κατεργασίας. Αν δεν κάνουμε την επιλογή αυτή, δεν μπορούμε να προσφέρουμε τίποτε στον κλάδο του χάλακτος. Και αυτή είναι η πρόταση που βλέπουμε τώρα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν δίνει δηλαδή σαφείς επιλογές και λύσεις. Αυτή είναι όλη η συζήτηση και αν θέλουμε να είμαστε σαφείς θα πρέπει ναι, να μην επανέλθουμε ως προς το 33% της δυνατότητας ε, για σύναψη συμβάσεων. Πολύ καλά, αυτό είναι απαραίτητο και πρέπει μάλιστα να δούμε αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε και υψηλότερα ποσοστά. Και δεύτερον, η φύση τη συμβάσεω σε σχέση με το θέμα των τιμών και θέτα από αυτά που λέει ο κύριο Ντε, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τον παραγωγό, μα από την διακύμανση των τιμών πρέπει να τον προστατεύουμε. Άρα θα πρέπει να έχουμε αρκετά μακρά περίοδο, μακριά περίοδο για να προστατεύσουμε ακριβώ τον παραγωγό. γιατί τις ποσοστές του γάλακτος, η κατάργησή τους, ό,τι και να λέμε, θα δημιουργήσει πολλές δυσκολίε στις περιοχές που ήδη βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση, σε δύσκολη κατάσταση και αυτό θα σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε λύσεις για να προστατέψουμε ε, τις περιοχές και του παραγωγού εκείνου που θα πληγούν από την κατάργηση των ποσοστών του 2015. Ο κύριο Μποβέ. Κοιτάξτε να σα πω θέλω και εγώ να πω ότι ο James έκανε ό,τι μπορούσε. Είχε ένα κακό κείμενο από την Επιτροπή ως βάση εκκίνησης. Δούλεψε όσο καλά μπορούσε. Αλλά είναι δύσκολο να κάνεις να βγάλεις ένα καλό αποτέλεσμα από κάτι που εξ αρχής είναι κακό. Και γιατί είναι κακό, γιατί η κατάσταση είναι καταστροφική σήμερα, από το 2009 και απανταχού δεν έχει αλλάξει τίποτα. Διαρκώς μειώνει το αριθμό των παραγωγών και δεν μιλάμε μόνο για μικρούς παραγωγούς ή μεσαίου μεγέθους παραγωγούς που εξαφανίζονται, ακόμη και μεγάλη παραγωγή με ναι. ένα ή δύο εκατομμύρια γάλα ποσοστώσει, ε, δύο εκατομμύρια τόνου γάλακτος σε ποσοστώσεις, βλέπουμε να εξαφανίζονται, διότι δεν μπορούν να διαθέσουν το προϊόν τους. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε διαρθρωτικά προβλήματα σήμερα. Και αυτό σημαίνει, αυτέ οι αναδιαρθρώσεις σημαίνουν ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση, ακόμη στην, και στην παραγωγή και ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα ε, διαδοχή στι ε, γεωργικέ εκμεταλλεύσεις, στι κοινοτροφικέ εκμεταλλεύσει, διότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα για ένα νέο να εξαγοράσει και να μπει στο επάγγελμα. Άρα τίποτα χειρότερα θα μπορούσαμε να κάνουμε από αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τι συστάσει τη. Οι συμβάσει ω διέξοδο από την κρίση. Όχι, δεν αποτελούν διέξοδο από την κρίση. Είναι συμβάσει οι οποίε εξυπηρετούν τη βιομηχανία και όχι τον παραγωγό. Ό,τι γίνεται, γίνεται για να προστατευτεί η παραγωγή, η βιομηχανία, η κατεργασία και όχι ο παραγωγό. Οι συμβάσει είναι ε, δεσμευτικές για τον παραγωγό, περιορίζουν τη δυνατότητα κινήσεώς του, τον δεσμεύουν υπερβολικά. Μάλιστα μέρο του κλάδου ούτε καν υφίσταται αυτόν τον περιορισμό και εδώ έχουμε να κάνουμε του συνεταιρισμού, αλλά εν πάση περιπτώσει μην κλείνουμε τα μάτια. στι πρώτες περιπτώσεις ο συνεταιρισμό μπορεί να είναι και χειρότερο από μια ιδιωτική επιχείρηση για τον παραγωγό και α μην ε, διακρίνουμε μεταξύ ιδιωτικού τομέα ή κλάδου και συνεταιρισμού. Πολλέ φορέ έχει ακόμη, χειρότερη ακόμη δυνατότητα πίεση βάρο του παραγωγού. Έτσι λοιπόν, Σημειώνω κλείνοντας ότι δεν θεωρώ αναπόδραστη την ε, κατάρριξη του συστήματος των ποσοστώσεων και πρέπει να επανεξετάσουμε στο σύνολο του το ζήτημα ε, πριν από το 2015. Πριν από το 2015. Και επίσης δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον παραγωγό εάν δεν έχουμε ε, διατίμηση και αν δεν έχουμε ε, στηρίξει την αυτή στο κόστο τη παραγωγή, υπέρ του παραγωγού, εάν δεν υπάρχει μια δυνατότητα να ε, απαλλάξουμε από την πίεση του ε, κλάδου της λιανικής και της μεταποίησης των παραγωγών και αν δεν ακολουθήσουμε αυτά τα οποία έχει ψηφίσει το Κοινοβούλιο μέσα στις νέες προτάσεις που θα υποβληθούν στο μέλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν μπορώ να πω παρά μόνο ότι ανησυχώ ιδιαίτερο ε, σήμερα για την κατάσταση και φοβούμαι ότι μπορεί η γνωμοδότηση αυτή του Κοινοβουλίου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τι ανισότητε μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και μεταποιητών. Καλώς, συνεχίζουμε κύριε Σέτμαν. Θα σας πω δύο πράγματα κι εγώ. Ξέρω ότι μερικοί εδώ μέσα θέλουν να έχουν τη δυνατότητα η παραγωγή να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν τα πράγματα είναι δύσκολα τότε θα δούμε ποιοι είναι οι πιστοί και ποιοι δεν είναι και ποιοι προσπαθούν δηλαδή να παίξουν διπλά παιχνίδια. Η αυγοβιομηχανία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που δυστυχώς οφείλεται σε αυτά που αποφασίσαμε εδώ μέσα αλλά δεν εξαρτάται και τόσο πολύ τελικά από την Ένωση. Τι έγινε εδώ πέρα. Αντί να μειωθούν οι τιμές μας δώσανε λέει διαχείριση της προσφοράς. Και εγώ θεωρώ ότι ο γαλακτοκομικός τομέας πρέπει να το πετύχει επιτέλους να δεχτεί την ε, πειθαρχία που απαιτείται και που αποφασίζουμε εδώ μέσα. γιατί εδώ βγάζουν από τη μήγα ξύγκη και από το σύστημα αυγά. Δεν θα καταφέρουμε αλλιώς ποτέ να ταΐσουμε όλο μας τον κόσμο και την αγορά. Κυρία Μαγκίνας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Από καταλαβαίνω έχουμε καθυστερήσει. Θα προσπαθήσω να ακριβώς Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση αυτή. Τώρα αυτό που προβλέπει τροπολογία 16 μπορούμε να το υποστηρίξουμε όμω με στην τροπολογία 29 ε, ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε λίγο περαιτέρω. Λεχθέντος αυτού θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο ότι αν οι συνεταιρισμοί δεν απαιτούν σύμβαση τότε θα εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη μέσα στη δομή να δουν οι συνεταιρισμοί το ισοζύγιο ε, προσφοράς και το κάτι ακόμα που το είπα και στους παραγωγούς, ε, πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων, επειδή μπορεί να αυξήσουν ε, την παραγωγή του γάλακτος, δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε και να το κάνουν. Οι ποσοστώσεις τους εμποδίσουν να το πράξουν και Προσπαθούμε εδώ να επανφεύρουμε ένα μηχανισμό για να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα με τις ποσοστώσεις χωρίς να ε, είναι τόσο αυστηρό το σύστημα. Δεν είμαι σίγουρη αν θα πετύχουμε το στόχο με τις συμβάσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη εδώ. Να πούμε στους παραγωγούς ότι υπάρχει κίνδυνος. Αν όλοι πιστεύουν ότι απλώς ε, επειδή άρονται ε, έρεται η μέγενη των ποσοστώσεων ότι μπορούν να παράξουν όσο θέλουν. Πρέπει να τους ε, προειδοποιήσουμε. Η δυσκολία για τους παραγωγού είναι ότι ακόμη και αν υπάρχει μείωση της ζήτηση, η τάση είναι να αυξάνεται η προσφορά γιατί πέφτουν οι τιμές και προσπαθούν να αυξήσουν ε, η παραγωγή την προσφορά και να διατηρήσουν αυτή τη λεπτή ισορροπία. Και θα πρέπει οι συμβάσεις να αποτελούν τμήμα της λύσης. Νομίζω ότι έχουμε την ευθύνη να μιλήσουμε με τους γαλακτοκόμους να ε, εξετάσουν το θέμα της ισορροπίας της αγοράς ανεξάρτητα από το αν ε, μιλάμε για συνεταιρισμούς ή όχι. Δίνεται πολύ έμφαση στη σχέση μεταξύ μεταποιητών και παραγωγών στην έκθεση. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε το σύνολο της ε, γαλακτοκομικής αλυσίδας μέχρι και το το εμπόριο. Δεν ξέρω πώ μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δίνεται υπερβολική έμφαση στην Κομισιόν για την ενδυνάμωση των ε, οργανώσεων παραγωγών. Ε, υπερχρησιμοποιείται στο στάδιο αυτό και δεν δίνεται τόση έμφαση στο ε, να δούμε τι συμβαίνει στο άλλο άκρο της αλυσίδας, ε, γιατί ε, δεν λέει κάποιος σας ε, μειώσουμε τη δύναμη ε, του τομέα του εμπορίου. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα αριθμίσουμε όλα αυτά, γιατί αν τελικά κάνουμε λάθος μπορεί να υπάρξει και άλλη μια κρίση στο γαλακτοκομικό τομέα και θα υπάρχει ζήτηση αν καταρρεύσουν οι τιμές ή καταρρεύσουν τα εισοδήματα ε, και θα ε, πρέπει να υπάρξει και θα υπάρχει υποστήριξη για τη λήψη μέτρων αγοράς. Υπάρχει εδώ ένα βήμα, γίνεται ένα βήμα προς την κατεύθυνση αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ε, σε σχέση ε, με το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουν οι παραγωγοί όταν θα εκλείψουν οι ποσοστώσει. Εγώ του λέω, κοιτάξτε, να είστε σίγουροι ότι η επέκταση θα σας ωφελήσει γιατί διαφορετικά θα υπάρξει τεράστιο κόστος που θα πρέπει να ή οι μεμονωμένοι παραγωγή. Έτσι λοιπόν ε, δεν ε, νομίζω ότι πρέπει εδώ να κάνουμε πολλές τροποποιήσεις, τροπολογίες, όμως ανησυχώ για τους συνεταιρισμούς ε, και έχουμε και το ξεχωριστό ζήτημα για το ποιος μπορεί να αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά για τα γαλακτοκομικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω για, θα αναφερθώ σε δύο προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί της Λετωνίας με, και που δεν θίγονται ακριβώς σε αυτό το έγγραφο. Καταρχήν ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί πολλές από τις τροπολογίες του είναι τελικά σαφέστερες από τις αρχικές προτάσεις της Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά. Για την 29 που αφορά τις συμβάσεις θα ήθελα να μιλήσω. Οι γεωργοί μας θεωρούν ότι καλύτερο θα ήταν τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν αν πρέπει να εφαρμοστεί υποχρεωτικά ή όχι αυτό το σύστημα των συμβάσεων, διότι στη χώρα μου έχουμε από το 8 και μετά την ε, συμφωνία που εφαρμόζεται για τα συμβόλαια και τις συμβάσεις και, που, και για όλες τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ παραγωγών και αγοραστών και με μεγάλη επιτυχία. Άλλο πρόβλημα που βλέπουν οι γεωργοί μας είναι ότι δίνονται διαφορετικοί αριθμοί 33%, 20%, 75% οι μικρότερες χώρες χρειάζονται μια εξαίρεση επειδή είναι μικρότερες και επειδή πρέπει να ανταγωνιστούν τις άλλες στην περιφερειακή τους αγορά. Η πρόταση του ορίου στο 75 που γίνεται στην έκθεση Νίκολσον στο σημείο 21 και 26.2 ή η τροπολογία 19 κατατίθεται για να δούμε με ποιους όρους μπορεί να χορηγηθεί αυτή η εξαίρεση. Δεν είναι σαφές πώς θα υπολογιστεί η παραγωγή αυτή σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή. Το, η πρόταση του 20% δεν μπορεί να γίνει δεκτή παρά μόνο εάν η προτινόμενη εξαίρεση εφαρμοστεί στις μικρότερες χώρες μέλη. Προς δεν το έχουμε επαρκώς εξετάσει, δεν είναι σαφές πώς μπορεί να εφαρμοστεί στη χώρα μου. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά σας παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομος. Yes, thank you, Mr. Chairman. I can see... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι προσελκύει το ενδιαφέρον αυτή η πρόταση. Αυτό δείχνει η συζήτηση. Τι είναι αυτό, Οπότε φαίνεται να μην καλύπτει όλε τι ανησυχίες και τα προβλήματα του τομέα των γαλακτοκομικών. Και βέβαια δεν ήταν καν αυτό η πρόθεσή μας. Δεν προσπαθήσαμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Ούτε και θα μπορούσαμε άλλωστε. Βεβαίω, ίσως θα πρέπει να μην λησμονούμε, όπως άλλωστε επισημάνθηκε, ότι κύριος παράγων της αγοράς είναι η αγορά, ε, της ε, κοινής γεωργικής πολιτικής είναι η αγορά. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ε, διασφαλιστικές δικλίδες, η δίκτυα ασφαλείας, με ρήτρε δηλαδή οι οποίες θα προστατεύουν τον παραγωγό σε μια περίπτωση ε, όπου λόγω της κατάρριξη των ποσοστώσεων αντιμετωπίζει δυσκολίε και χρειάζεται μια επιπλέον ενίσχυση στην διαπραγματευτική του ισχύ για να μπορέσει να επιβιώσει, αλλά δεν είναι αυτό αποκλειστική λύση. Πάντω αυτό είναι το επίκεντρο ε, των μελημάτων μα, ότι δηλαδή με την κατάρριξη των ποσοστώσεων αποδυναμώνεται ο παραγωγό στην πραγματευτική του ισχύ και κυρίω σε σχέση με τι μονάδε με τις μονάδες επεξεργασίας γάλακτος, ε, Για δε την θέση του μεμονωμένου παραγωγού μέσα στο συνεταιρισμό θεωρώ ότι είναι σφάλμα του παραγωγού του ίδιου εάν δεν έχει αρκετά ισχυρή φωνή μέσα στο συνεταιρισμό του. Πρέπει ο ίδιος να μεριμνήσει ώστε να επιλέγει πρόσωπα και διοίκηση στο συνεταιρισμό που να ε, καθιστούν ε, δυνατή τη συμμετοχή τους σε αυτά που να μην τον αποκλείουν. Επίσης, η πρότασή μας στο στόχο έχει για κάποιον που δεν είναι μέλος συνεταιρισμού και κυρίως γι' αυτόν να αναπτύξει μια οργάνωση ή να συμμετάσχει σε μια οργάνωση παραγωγών κατ' εξαίρεση των κανόνων περί ανταγωνισμού που θα μπορεί να διαπραγματευτεί αποκλειστικά ε, και μόνο τις τιμές. Κατά αποκλειστικότητα και μόνο τις τιμές. Ναι. Κατά το οποίο δεν επέτρεπε μέχρι τώρα η όρη του δικαίου του ανταγωνισμού. Αυτό το επιτρέπουμε τώρα γιατί βλέπουμε ότι κερδίζουμε σε αποτελεσματικότητα όχι μόνο στον χώρο του, των γαλακτοκομικών αλλά για ολόκληρη την κοινωνία. Και έτσι αυτό, αυτή η συμμετοχή σε μια οργάνωση παρακοχών είναι το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή σε ένα συνεταιρισμό γιατί μπορεί ο, ο παρακοχός και γι' αυτό έχουμε και συγκεκριμένο χρονικό όριο, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να συμμετάσχει σε μια οργάνωση, όχι μόνο με αυτό σκοπό αυτή τη συμμετοχή, αλλά προκειμένου να ενθαρρύνουμε και να ενθαρρύνουμε την οργάνωση αυτοπεραγωγών να μετατραπεί στη συνέχεια σε ένα συνεταιρισμό, αλλά και να ε, προχωρήσει σε ανάπτυξη των δομών και υποδομών της, ακόμη και με εξοπλισμό τύπου φορτηγών ε, ή γεωργικών μηχανημάτων άλλων, που θα τις επιτρέψουν να αναπτύξει τα στερεότητες της περισσότερο. Και αυτό επίσης δεν ήθελα να επισημαίνω ότι δεν ε, ε, αποτελεί πάντοτε επιβάρυνση ως προς την τιμή γάλακτος για τον παραγωγή, του γάλακτος για τον παραγωγό, διότι ακούστηκε νωρίτερα ότι διαρκώς θα πιέζεται προς τα κάτω η τιμή του γάλακτος. Αυτό μπορεί να ισχύει για κάποιον ο οποίος ασχολείται μόνο με την παραγωγή αποκλειστικά και μόνο ε, γαλακτοκομικών προς κατανάλωση παραδοσιακού τύπου, δηλαδή γάλα, βούτυρο ε, και ούτω καθεξής. Αλλά θα πρέπει τώρα ε, να κοιτάξουμε και την άλλη εκδοχή. Μια μονάδα επεξεργασίας γάλακτος θα πρέπει να κοιτάει τον στόχο της βελτίωσης προσθέμενης αξίας, όχι μόνο δηλαδή να εξασφαλίσει καλύτερες ε, τιμές για τον παραγωγό της, αλλά περισσότερο κέρδος για τον παραγωγό. Άρα είναι διαφορετική η κατάσταση των παραδοσιακών λεγόμενων γαλακτοκομείων που, που περιορίζονται στην ε, στόχευσή τους στα παραδοσιακά προϊόντα και εκείνων τα οποία είναι πιο καινοτόμα και αναζητούν νέες λύσεις. Και υπόθηκε σαν ποσοστό το 33% σε ρεαλιστική μάλιστα εξισορρόπηση μεταξύ των αναγκών ε, για τις ανάγκες για ε, καλή διαπραγματευτική ισχύ, ικανοποιητική διαπραγματευτική ισχύ για τον παραγωγό, αλλά χωρίς βέβαια να, το, επιτρέπεται στις οργανώσεις των παραγωγών να εξασφαλίσουν ε, μονοπωλιακή ή ιονίμιο μονοπωλιακή θέση και πάνω απ' όλα να μην συμπιέσουν το μικρό και μεσαίο παραγωγό. Αυτή είναι η πρότασή μα και έχουμε και διασφαλιστική δικλίδα ω προ τον ανταγωνισμό, μέτρο το οποίο θεωρούμε θετικό, διότι εν γέννη ο παραγωγό και ο ιδιαίτερο παραγωγό γάλακτο μπορεί να είναι ε, σε ασθενέστερη θέση, αλλά εάν συνεργαστούν πολλοί παραγωγοί μαζί, μπορεί εν σχέση με μια μονάδα επεξεργασία γάλακτο, μάλλον μικρού μεγέθου, να είναι πολύ ισχυρότερη, να έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ και ειδικό βάρος. Αυτό λοιπόν ως ασφαλιστική δικλίδα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Επιμένουμε επίσης ότι θα πρέπει να γίνεται ε, ελεύθερα και απεριόριστα η διαπραγμάτευση των όρων τη συμβάσεω χωρί χρονικά όρια, χωρί μέγιστα ή ελάχιστα χρονικά όρια, χωρί συμμετοχή των κρατών μελών που θα μπορούσαν ενδεχομένω να επιβάλλουν ανώτατο ή κατώτατο όριο διάρκεια αυτή τη σύμβαση. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι ελεύθεροι όροι που θα διαπραγματευτούν τα μέρη. Και αυτό γιατί, διότι θα μπορούσαμε στη μία περίπτωση να ενισχύσουμε τη θέση του ε, αγοραστή ή σε μια αντίστροφη περίπτωση του πολιτή. Γι' αυτό θέλουμε να είναι τελείως ουδέτερες αυτές οι συμβάσεις. Και επίσης θα θέλαμε να παρέμβουμε κατά τρόπον την στου στους κανόνες των συνεταιρισμών, που είναι πολύ διαφορετικοί κανόνες, γιατί υπάρχουν κάποιοι συνεταιρισμοί που λένε ότι μπορεί κανείς να γίνει μέλος μόνο εάν δίνει 100% της παραγωγής του σε αυτόν, ενώ κάποιοι άλλοι ως όρο συμμετοχής έχουν ε, ένα ποσοστό μόνο ε, πώληση ε, των προϊόντων ε, στον συνεταιρισμό. Δηλαδή αφήνει τον παραγωγό ελεύθερο να διαθέτει το προϊόν του και σε κάποιον άλλον. Ε, αυτό λοιπόν πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να το χειριστούμε. Και μπορεί μέλο συνεταιρισμού να επιλέξει να οργανωθεί μέσα σε μια οργάνωση παραγωγών που θα διαπραγματευτεί στη συνέχεια με τον συνεταιρισμό ή με μια μονάδα κατεργασίας γάλακτος υπό τον όρο ότι δεν αποκλείεται αυτό από τους όρους συμμετοχής στον συνεταιρισμό. Όλα αυτά όμως τα επισημαίνω δηλώνοντα ταυτόχρονα ότι δεν προσπαθούμε να εφεύγουμε νέου κανόνε, ούτε επιτρέπεται να βγάλουμε νέου κανόνε που θα παρεμβαίνουν στην απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των κανονισμών, των ε, συνεταιρισμών, που σε τελευταία ανάλυση έχουν ορίσει με την ομοθεσία του τα κράτη-μέλη. Οι Βρυξέλλε δεν πρέπει να παρέμβουν σε αυτό το επίπεδο. Και επίση θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όντω, και συμφωνώ σε έναν βαθμό, ε, τα προβλήματα εντοπίζονται στον ε, τομέα τη λιανική. Αλλά ο παραγωγός γαλακτός δεν διαπραγματεύεται με τον λιανέμπορο. Διαπραγματεύεται είτε με τον συνεταιρισμό του, εφόσον υπάρχει δυνατότητα διαπραγματεύσει, είτε με την επιχείρηση, την μεμονωμένη επιχείρηση επεξεργασία κράτου. Εάν λοιπόν ο συνεταιρισμό κάνει σωστά τη δουλειά του, εάν ο συνεταιρισμό εξασφαλίζει καλή τιμή, ικανοποιητική τιμή για τον παραγωγό, ορθή τιμή, είναι η καλύτερη λύση αυτή. Έτσι βρίσκουμε τη σωστή ε, τιμή για τον παραγωγό όχι με μια ελάχιστη τιμή που θα επιβάλαμε ή με τον έλεγχο των όγκων ε, που θα πολλούνται και ούτω καθεξής. Δεν είναι αυτός τρόπος να εξασφαλιστεί μεγαλύτερο μερίδιο από την αξία της αλυσίδας ε, ε, διάθεση του γάλακτος για τον παραγωγό. Επαναλαμβάνω λοιπόν και υπογραμμίζω ότι πρόκειται για ένα βήμα, μόνο ένα βήμα, όμω, στον στόχο τη ενίσχυση τη διαπραγματευτική ισχύω του παραγωγού, χωρί να αποτελεί πανάκια, και ε, μαγική λύση και επίσης προφανές είναι ότι δεδομένων των ε, συγκρούσεων απόψεων, των ε, αντικρουμένων απόψεων που διαπιστώνονται εδώ, τέτοιου είδους προτάσεις δεν θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ούτε στο Κοινοβούλιο ούτε και σε επίπεδο Συμβουλίου συνένεση. Πολλά θα είχα να πω ακόμη, Πρόεδρε, για το παρατηρείο τιμών, για τις εξουσιοδότηση πράξεις, το μάξιο της πενταετίας, και πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν είναι η ώρα νομίζω. Θα σταματήσω εδώ, καλώντας τους ε, κυρίους βουλευτές να καταθέσουν τις τροπολογίες, τις οποίες θα εξετάσουμε και πέραν αυτού του σταδίου θα μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Και τώρα ο κύριος Νίκολσον. Uh, Uh, thank you very much. Αλλάζουμε επίτροπο, αλλά όχι υπαλλήλου τη Κομισιόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να του ευχαριστήσω όλου όσου πήραν το λόγο. Ξέρω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον για πολλού από του συναδέλφου, αλλά ακόμη και η δική μου πεποίθηση μάλλον δεν ανταποκρίθηκε στην πραγματικότητα. Φαίνεται πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για πολλού συναδέλφου και πολλέ περιοχέ στην Ευρώπη. Σας ε, ευχαριστώ κύριε Μποβέ για όσα είπατε, γιατί πραγματικά ε, με απαλλάσσετε αν κάποιος νομίζει ότι έκανα κακή δουλειά. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει νόημα να ε, Έχουμε τώρα περαιτέρω συζήτηση, θα το δούμε αυτό βάσει των τροπολογιών που θα κατατεθούν και με τους σκιώδεις ηγητές θα προσπαθήσω να καταλήξουμε σε μια συνένεση και όπως είπε και η Κομισιόν αναγνωρίζω ότι ενώ λέω 20% δεν θα αρκέσει το 20% αλλά θα πραγματευτούμε για να δούμε ε, ποιο θα είναι μια λογική λύση, αν θα πρέπει να έχουμε 33% ή κάτι άλλο. Ο κύριος Δαντέ ε, είπε ότι πρέπει να, παρα, να παρακολουθούμε την αγορά με σταθερό τρόπο, ενώ άλλη είπε να, αν το ξανακάνουμε αυτό λάθος θα είναι πλήρης καταστροφή για όλους τους παραγωγούς, τους μεταπηδές κτλ. Και η Μαρία είπε και εγώ είπα ότι είναι ατελής η έκθεση γιατί δεν ε, υπάρχει εδώ το λιανεμπόριο, δεν υπάρχουν οι λιανέμποροι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ε, νομοθετούμε για δύο τμήματα της ελισίδας όταν αφήνεται εκτός ένα άλλο τμήμα της ελισίδας. Όμως μάλλον αυτό θα το δούμε πιο μακροπρόθεσμα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η αστάθεια των τιμών. Ε, γιατί κοιτάξτε, αν ε, έχουν ε, παραδείγματο χάρη υπογράψει μια σύμβαση η παραγωγή πριν 9-12 μήνες, τότε δεν είναι και πολύ σχετικό και αυτό το συμβόλαιο σήμερα, επειδή έχουν αυξηθεί οι τιμές και στα λοιπάσματα και στα καύσιμα και στις ζωοτροφές. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα βαθμό ευελιξία. Πρέπει να υπάρχει ευελιξία και από την πλευρά των παραγωγών αλλά και των μεταποιητών. Και ε, σήμερα αυτή η αστάθεια στην παγκόσμια αγορά είναι, ε, μας δείχνει πόσο δύσκολο είναι για όλους μας να δούμε ποιο είναι ο ορθό δρόμο προ τα μπρο. Και συμφωνώ με τον εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Νομίζω ότι ο καλύτερο τρόπο να δούμε την πρόταση αυτή είναι ότι αυτό είναι ένα βήμα σε ένα μακρύ δρόμο και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Πρέπει να δούμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Κοιτάξτε, μία σύμβαση είναι ένα που μαχαίρι Δηλαδή λειτουργεί για τον παραγωγό αλλά και για τον μεταποιητή. Αν αυξηθεί η τιμή ή μειωθεί η τιμή, τότε πρέπει να ε, πληρωθούν οι ώρες της σύμβασης. Δεν μπορεί να πει ο παραγωγός να σου δίνω νέο γάλα, ούτε ο μεταπητής μπορεί να πει δεν παίρνω το γάλα σου. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να βρούμε που είναι η ευελιξία και του συμβιβασμούς που χρειάζεται αν αυξομοιωθούν οι τιμές. Πρόεδρε, ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος γιατί ξεφύγαμε, αλλά θα πω κάτι ακόμα. το που ακούστηκε εδώ σήμερα. Η Ευρώπη έχει 27 κράτη-μέλη, μέχρι την εφαρμογή μάλλον θα 29. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές περιφέρειες, περιοχές και υπάρχουν και πολλές διαφοροποιήσεις και στο εταιρικό ενός κράτους μέλους και ένα θα τον κάνει για όλους. Και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και το έχω και περισσότερο κατά νου όταν μιλάμε για την ευελιξία. Έτσι λοιπόν τα κρατημέλη πρέπει να έχουν την ευελιξία να καλύψουν τις ανάγκες των δικών τους περιφερειών. Είναι τόσο απλό, δεν θα είναι εύκολο, αλλά περιμένω τι τροπολογίε σας και αναμένω να συνεργαστώ μαζί σας και να ξαναβρούμε ένα συμβιβασμό που χρειάζεται. Ελπίζω να μπορέσουμε να να παρουσιάσουμε κάτι και κατάλαβα ότι θα έπρεπε να βάλουμε μία ρήτρα ραντεβού, μία ρήτρα επαναθεώρησης, να το ξαναδούμε μετά από δύο μισή έτη, γιατί δεν νομίζω ότι ε, όλα θα τα κάνουμε σωστά τελικά έτσι με την πρώτη απόπειρα και μάλλον θα πρέπει να επανέλθουμε για να ξανασυζητήσουμε την Κομισιόν σε μετέπειτα στάδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ καλή η συζήτηση για το γαλακτοκομικό τομέα και ας προσπαθήσουμε τις επόμενες εβδομάδες ε, να καταλήξουμε στους απαραίτητους συμβιβασμούς. Ευχαριστώ. Η κατάθεση τροπολογιών έως τι 22 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Σας υπενθυμίζω. Και έτσι περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερικής διάταξης που είναι το εργαστήριο για την ε, ποιότητα για τα στήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα. Έχουμε δύο προτάσει ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη ρυθμίση των συστημάτων ποιότητας το ένα και το άλλο για τα πρότυπα εμπορίας. Είναι προτάσεις ε, που έχουν ε, λάβει υπόψη πολλές από τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Έχουμε έκθεση του κυρίου Σκοτά και σήμερα θα γίνει συζήτηση στο workshop μας όπου καλωσορίζω τους ειδικούς Ντένις Παντίνη, τον κύριο Παντίνη, ο οποίος θα μιλήσει για την πολιτική ποιότητα ε, από το 2013 και μετά, και τον κύριο Ζιλ Αλέχ, ο οποίος θα μιλήσει για τις τοπικές αγορές και τις ε, μικρότερους παραγωγούς. Ο κύριος Παντίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Noi eh, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γεωργίας ε, Αγροτική Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου που με κάλεσε σήμερα να μιλήσω σε αυτό το εργαστήριο για το μέλλον ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής Ποιότητα. Ε, θα παρουσιάσω κατευθείαν την εκθεσή μου που θα εστιαστεί σε τρία κυρία σημεία. Καταρχήν, θα περιγράψω ποιος είναι ο οικονομικός ρόλος των προϊόντων ποιότητας ε, στο αγροπεριστατιστικό πλαίσιο της Ευρώπης και ποιες προβληματικές ενδιαφέρουν τους παραγωγούς. Το δεύτερο τμήμα ε, θα είναι να κατανοήσουμε ποιες είναι οι απαντήσεις σε αυτές τις προβληματικές των παραγωγών και για να κλείσουμε ορισμένε παρατηρήσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και τις οικονομικές αξίες αυτών των προϊόντων. Καταρχήν, το πρώτο σημείο το οποίο θέλω να σας επισημάνω είναι ότι η πολιτική ποιότητα σίγουρα έχει, υποδεχθεί, έχει γίνει ε, αποδεκτή από τους ευρωπαϊκούς παραγωγούς γιατί μέχρι σήμερα από το 2002 έχουμε ε, εγγράψει δεκτές προϊόντα προστευόμενης γεωγραφικής προέλευσης και προστευόμενης γεωγραφικής ε, ένδειξης. Αυτό δεν οδήγησε σε σημαντική ε, ανταπόκριση από τους καταναλωτές. Ε, μόνο το 8% του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα διάφορα σήματα προστατευόμενης γεωγραφικής προέλευσης και pop. Ε, στην Ιταλία ή στην Πορτογαλία είδαμε κάποια διαφορετικά αποτελέσματα και βέβαια ε, αν δείτε τα στοιχεία της διαφάνειας θα δείτε ότι τα τελευταία τέσσερα έτη από το 2005 στο 2008 ε, έναντι μίας αύξησης 15% των εγγραφών η αξία των προϊόντων ε, αυτών αυξήθηκε μόνο 6% για να κατανοήσουμε καλύτερα τι σημαίνουν αυτά τα προϊόντα. Ε, έχουμε 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ και ε, τις αξίες αυτών των προϊόντων και είναι μια αξία κατώτερη από ε, τα έσοδα της πρώτης επιχείρησης τροφίμων και αναψυκτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτω του 2% από τι εξαρτάται ε, το πρόβλημα σχετίζεται με το ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός κατακαιρματισμένου παραγωγικού συστήματος, μικρή παραγωγή και μεταπιτές που παράγουν μικρές ποσότητες. Ε, είναι μιας μέσος υπολογισμός μας λέει ότι έχουμε αξία κάτω του 20, 20.000 ευρώ. Στο εσωτερικό αυτού του συστήματος βέβαια υπάρχουν και άλλες συνιστώσεις όπως της μπύρας ή των τυριών ή των προπερσκευασμένων κρεάτων όπου έχουμε ε, μεγαλύτερα αριθμητικά στοιχεία παραγωγής ε, η αξία μεγαλυτερα ρυθμιτικά στοιχεια παραγωγης η αξια φτανει ε, στο 55% ε, των προϊόντων αυτών, ε, των προϊόντων ποιότητας, αν και έχουμε μόνο 35% στις εγγραφές. Και βάση αυτής της έλλειψης ανάπτυξης είναι το ότι δεν έχει επαρκή γνώση ο καταναλωτής για αυτά τα σήματα. Γιατί ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονό ότι όταν ο καταναλωτή το αναγνωρίζει, είναι διατεθειμένος να πληρώσει περισσότερο. Και αυτό το βλέπουμε για τι κυρίε κατηγορίε, όπου βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο τα προϊόντα ποιότητα στην αγορά έχουν πιο υψηλέ τιμέ ε, από όλο το μέσο όρο των προϊόντων. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε γιατί έχει να κάνει και με τους στόχους ε, ε, της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ είναι το ότι τα προϊόντα ε, ποιότητας κατορθώνουν να εκφράσουν μια καλύτερη ικανότητα παραγωγής δημοσίου αγαθού. Συνδέονται ε, με την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και υπάρχουν και κάποιες οικονομικές συνέργειες ε, που τίθεται ε, σε εφαρμογή και μάλλον μίσο όπως του τουρισμού λόγου χάρη. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου. Ποιες είναι οι ανάγκες που η παραγωγή των προϊόντων ποιότητα εκφράζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουν να βελτιώσουν την αγωνιστικότητά του και τη θέση του. Μία από τι πρώτε ανάγκε σχετίζεται με την διεθνή προστασία. Το 18% τη αξία των προϊόντων ποιότητα ε, εκτό ε, τη εθνική αγορά όπου παράγονται και αυτό το 18% πετυχαίνεται στις αγορές τρίτων χωρών. Αυτή η τιμή δεν είναι πολύ ψηλή, αλλά ε, δείχνει ποια είναι η δυναμική της αγοράς, ε, που είναι σίγουρα ανώτερη. Και αυτό συμπεραίνεται από το γεγονός ότι στο πλαίσιο πολλών τρίτων χωρών ε, υπάρχουν μεταναστευτικά φαινόμενα τέτοια παραγωγή. Μία μελέτη που έγινε πέρσι μα έδειξε ότι στην αγορά των ΗΠΑ η ποσόστοση των προϊόντων προϊόντων ε, που ε, είναι απομίμηση ιταλικών προϊόντων ποιότητας ε, είναι παρόμοιες με τα αληθινά και αυτό μας δείχνει ποια είναι η δυναμική της αγοράς για αυτά τα προϊόντα. Τι προτείνει το πακέτο είδες μέτρων ποιότητα για να λυθεί αυτό το, αυτή η προβληματική. Σίγουρα ενισχύει την προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο χάρη στο ότι προτείνει τη δημιουργία συστημάτων προστασίας, προστευόμενης ε, ονομασία πρόελευση και προστευόμενης γεωγραφική ένδειξη σε όλα τα κράτη-μέλη. Και ε, ε, Επίσης, προβλέπεται η χρηματοδότηση των απαραίτητων δραστηριοτήτων για να τεθούν σε εφαρμογή όλες οι δραστηριότητες υπεράσπισης από παράνομη χρήση ε, έτσι λοιπόν, των σημάτων αυτών, έτσι λοιπόν ε, υποστηρίζονται οικονομικά οι απαραίτητε δραστηριότητε για να αποφευχθούν να υπάρχουν φαινόμενα που μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση στον καταναλωτή μεταξύ αληθινών και ψεύτικων σημάτων ε, POP. Όμως το πρόβλημα παραμένει σε διεθνές επίπεδο όπου η προστασία που δίνει ο κανονισμός του 2006 δεν ισχύει. Έτσι λοιπόν ε, εδώ δίνεται μία υποστήριξη από τη Συμφωνία Τρίψη για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Μια πιθανή βοήθεια εγγράφεται στο πλαίσιο του άρθρου 23 της συμφωνίας αυτής, όπου ήδη το 2004 δηλωνόταν η βούληση να υπάρχει μια πολυμερής, ε, ένα πολυμερές μητρό για να διευκολύνουμε ε, την προστασία της ονομασίας προέλευσης των ίνων. Όμως ε, ποτέ στο πλαίσιο αυτό δεν καθορίστηκε ποιοι τρόποι πρέπει να ακολουθηθούν για να δημιουργηθεί το μητρό και σε ποιο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, ε, είδαμε να υπάρχουν ε, διάφορες θέσεις ε, από την πλευρά του Παγκόσμιου Οργανισμού Ίνου και Αμπέλου. Ε, όμως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την υποστήριξη και άλλων χωρών όπως Ελβετία, Τουρκία, ε, χωρίς από την Αφρική και Βραζιλία στην επέκταση αυτού του μητρώου όχι μόνο στους ίνους αλλά και στα άλλα διατροφικά προϊόντα. Θα πρόκειται για ένα μητρό υπό τη διαχείριση της γραμματείας του ΟΗΒΕ που θα ήταν δεσμευτικό και ε, όταν θα είχε εγγραφεί η ονομασία προέλευσης θα αποτελούσε απόδειξη ε, ότι υπάρχει συγκεκριμένη σύνδεση με, το συγκεκριμένη, με τη συγκεκριμένη επικράτεια. Όμως έχουμε άλλες χώρες όπως Αυστραλία ή Πακαναδάς και Νέα Ζηλανδία που αντιθέτως δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να επεκταθεί αυτό το μητρό ε, στα τροφικά προϊόντα εκτός των ίνων και θέλουν ε, μάλιστα να μην συμπεριλαμβάνεται ε, ένα δεσμευτικό σύστημα ε, για τις χώρες που δεν συμμετέχουν. Τώρα, οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Ίνου και Αμπέλου περιλαμβάνει ορισμένα βήματα που πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε στον καθορισμό του Μητρώου. Δηλαδή, πώς πρέπει να γίνεται η κοινοποίηση, γραφή και οι νομικές συνέπειες ε, που προκύπτουν. Και για να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσει αυτέ, η δέσμη μέτρων για την ποιότητα προσπαθεί να ευθυγραμμίσει τον ορισμό των νομασιών προέλευση και των προστατευμένων γεωγραφικών ενδείξεων με αυτά που έχουμε σε διεθνέ επίπεδο. Εν τω μεταξύ, για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ε, κάτι ε, ακόμη χρήσιμο για την προστασία των ομισιών αυτών θα ήταν να υπάρξουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ περιφερειών και ομάδων χωρών προκειμένου ε, αυτές οι συμφωνίες να δεσμεύουν εν λόγω μέρη. κάθε φορά όμως θα είχαμε επανάληψη αυτών των συμφωνιών. Επειδή δεσμεύονται μόνο τα συγκεκριμένα μέρη. Τώρα, μία άλλη απέτηση που αναφέρθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση είναι το θέμα της ενίσχυσης της ε, δεσμευτική, της ε, ισχύω ε, της, της σύναψης συμβάσεων. Καταρχήν πρέπει να μιλήσουμε αυτό λόγω του ότι υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να, μάλλον το ότι έχουμε ε, πολλές μικρές επιχειρήσεις ε, όπου κάθε μία παράγει μικρές ποσότητες προϊόντων. Ε, ε, βλέπετε στη διαφάνεια ορισμένα παραδείγματα. Φαίνεται ότι στην Ιταλία, παραδείγματο χάρη, έχουμε ε, παραγωγή πάνω από ένα εκατομμύριο τόνων και έχουμε 76.000 εκμεταλλεύσεις, ενώ στη Γαλλία έχουμε 56.000 ε, εκμεταλλεύσεις για 600.000 τόνους ε, προϊόντων. Mm. Όμως, ε, αν δούμε για τα τυριά, έχουμε στην Ιταλία 450.000 τόνους και έχουμε 1.400 εκμεταλλεύσεις, ενώ στην Ισπανία έχουμε ακόμα μεγαλύτερο κερματισμό. 29.500 τόνοι από 433 εκμεταλλεύσεις. Τώρα, το πρόβλημα συνδέεται με το ότι αυτή η μικρή παραγωγή περνούν μέσω από τους μεγάλες επιχειρήσεις της διανομής και περνούν το σχάρι τα γαλλικά τυριά πολλούνται μέσω από ε, αυτού, αυτές τις επιχειρήσεις και μιλάμε στην Ιταλία για το 65% των όγκων παραγωγής ε, και η παραγωγή των ε, σημάτων των μαρκών ποιότητας ε, ε, ουσιαστικά ε, είναι αντιμέτωποι με το εξή. Βλέπετε στη διαφάνεια ότι 13,7 εκατομμύρια παραγωγών για να μπορέσουν να φτάσουν σε μία αγορά 55 εκατομμύρια ε, συγγνώμη, 550 εκατομμυρίων πρέπει να περάσουν από συμπληγάδες, ε, δηλαδή πρέπει να περάσουν από του, τις επιχειρήσεις μεγάλης διανομής. Αυτό οφείλεται στο ότι οι επιχειρήσεις, ε, τις μεγάλες επιχειρήσεις διανομής παρουσιάζουν ισχυρή συγκέντρωση στην αγορά. Στη Γαλλία οι πέντε πρώτες αλυσίδες διανομής συγκεντρώνουν ε, περίπου το 80%, στη Γερμανία έχουμε το 71%, στην Ισπανία το 48% και στην Ιταλία το 27%. Τώρα, αν αυτό αποτελεί πρόβλημα για όλους τους παραγωγούς στην Ευρώπη, ε, στην περίπτωση που έχουμε παραγωγούς ε, προϊόντων ποιότητας είναι πιο έντονο το πρόβλημα για μια σειρά λόγων. Καταρχήν γιατί ε, καθίσταται ομογενοποιημένες όλες οι παραγωγές από τους διάφορους παραγωγούς και δεν επιτρέπεται στους παραγωγούς αυτούς να έχουν τους πόρους για να προωθήσουν τη δική τους μάρκα. Αυτό σημαίνει ότι στην ε, περίπτωση που έχουμε υψηλούς όγκους παραγωγής που προέρχονται από τόσους πολλούς μικρούς παραγωγούς, όταν έχουμε συγκέντρωση ε, στη διανομή, το ε, αποτέλεσμα της πτώσης των τιμών αφορά το σύνολο των παραγωγών των προϊόντων ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχουμε αστάθεια των τιμών και πτώση των τιμών, και μάλιστα και κάτω από το κόστος παραγωγής ο μονομένος παραγωγός δεν μπορεί να μειώσει το ίδιο του το κόστος γιατί δεσμεύεται πω την ομοθεσία για την παραγωγή. Έτσι λοιπόν πρέπει να υποστεί αυτή τη ζημία και συσσωρεύει αυτή τη ζημία και σημαίνει ότι τελικά πρέπει να καταλήξει στο να κλείσει την επιχείρηση που παράγει αυτό το προϊόν και υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος ε, στις πτυχές που αναφέραμε προηγουμένω, δηλαδή στη δημιουργία, στην παραγωγή δημόσιων αγαθών, ε, στην ε, στο κλείσιμο των επιχειρήσεων, ε, ανεργία κτλ. Τι κάνει τώρα η δέσμη των μέτρων ποιότητα για να βελτιώσει την κατάσταση. Αφενός αναγνωρίζει το ρόλο και την ευθύνη των ομίλων ε, όπως οι ενώσει παραγωγών στην δραστηριότητα που έχει ως στόχο να κοινοποιήσει στον καταναλωτή σε τι διαφέρουν τα προϊόντα αυτά σε σχέση με τα άλλα. Αλλά βεβαίως για να βελτιωθεί η συμβατική ισχύ αυτών των παραγωγών θα ήταν καλύτερο να μπορέσουμε να σκεφτούμε με όρους προγραμματισμού της παραγωγής σε μια οπτική βελτίωση της ποιότητας ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς. Μία τελευταία πτυχή που θέλω να καταδείξω και αποτελεί μία ε, εγκάρσια απέτηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Γεωργία και που αναφέρεται ε, και στην ΕΑΠΑΚ είναι το θέμα της ε, μείωσης της γραφειοκρατίας. Το πακέτο για την ποιότητα εισαγάγει τρόποποίησης προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η απλούσταση μειώνοντας το χρόνο για την ανάλυση των αιτήσεων, για την εγγραφή των προϊόντων POP και προστευμένων γεωγραφικών ενδείξεων από τον ένα χρόνο στους 6 μήνες. Όμως, ε, δια διαφοροποιείται, εξακολουθεί να παραμένει διαφοροποιημένο το καθεστώς και το μητρό για τα κρασιά και για τα διατροφικά προϊόντα. Ε, θα μπορούσαμε, παραδείγματο χούμε, ε, να έχουμε συνέργειες στην περίπτωση αυτή όταν έχουμε εκστρατείες πρόθεση των προϊόντων αυτών. Μία άλλη πτυχή που αναφέρεται πολλάκι ε, στην πρόταση κανονισμού είναι αυτό της χρήσης των καταξουσιώτων της πράξεων. Όπως ξέρετε, το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η Κομισιόν έχει την ε, αρμοδιότητα, την εξουσία μέσω των ε, πράξεων αυτών, την καταξιοδότηση να να χρησιμοποιήσει αυτές τις πράξεις για να ε, περιλάβει στην νομοθετική πράξη μη ουσιαστικά στοιχεία εισαγάγοντας ή προσδιορίζοντας κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά ή εισαγάγοντας κάποια νέα στοιχεία στην νομοθετική πράξη. αυτή ε, η πρακτική θα έπρεπε να μην ε, αποτελεί συχνή χρήση, θα έπρεπε να αποτελεί εξαίρεση ε, για να μην διακυβευτεί η αρχή της διαφάνειας των ίδιων των δημοθετικών διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, με όλες αυτές τις σκέψεις πρέπει να έχετε κατά νου ότι η πρόταση κανονισμού για τα καθεστώτα ποιότητας, η διαδικασία των κατεξουσιοδότηση πράξεων εμφανίστηκε σε 18 άρθρα από τα 51 mm. και σε πολλές περιπτώσεις ε, προσδιορίζονται και στοιχεία που, είναι, που δεν είναι δευτερού σημασία. Δηλαδή, όταν μπορούμε να καθορίσουμε ποια προϊόντα θα μπορούσαν να τη χάνουν αυτού του καθεστώτο ε, ή παραδείγματο χάρη να ε, ρυθμίζονται ορισμένε παρεκκλήσει. Και φτάνω τώρα στα συμπεράσματα με κάποιες ε, παρατηρήσεις προσωπικού χαρακτήρα. Εγώ πιστεύω ότι ε, η σχετικότητα και η ισχύ ενό γεωπιστητιστικού συστήματο ποιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στον αριθμό των εγγραφών, αλλά στην κοινωνικο-οικονομική αξία που εκπροσωπούν αυτά τα προϊόντα όπως και για όλα τα άλλα γεωπιτιστικά προϊόντα και για τα προϊόντα αυτά, εγκυμένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα ή προϊόντα pop, θα μπορούσαμε να ε, δούμε πόσο εισόδημα μπορούν να παράξουν για τον παραγωγό και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε δηλαδή τη δική τους ανταγωνιστικότητα στην αγορά. Πολλά από αυτά τα προϊόντα έχουν περιορισμένες ε, δυνατότητες, ε, ε, όμως ε, πολλές φορές το πρόβλημα που συναντάνε είναι το πρόβλημα της πρόσβασης στην αγορά και ακριβώς γι' αυτό μία από τις κύριες αδυναμίες της ευρωπαϊκής πολιτικής ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί το εξή. Ότι πέρα από το να αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα ή η αξία των προϊόντων αυτών, ε, πρέπει να τίνει να τα διατηρήσει αυτά τα προϊόντα. Αλλά αν ε, έχουμε μια πολιτική που απλώ ε, μιλά για τη συντήρηση και όχι για την ανάπτυξη, μιλάμε για κοινωνική πολιτική και όχι για οικονομική πολιτική. Έτσι λοιπόν το σημαντικό εδώ είναι να θεωρήσουμε ότι για να βελτιώσουμε αυτή την πολιτική εμείς δεν θα έπρεπε ε, να στοχεύουμε στην αύξηση του αριθμού των κατεχωρήσεων, δηλαδή σε 10 χρόνια να έχουμε 2.000, 3.000 τέτοια προϊόντα θα ήταν καλύτερο να προσπαθήσουμε να διπλασιάσουμε την οικονομική αξία των χίλιων καταχωρήσεων που έχουμε σήμερα. Και για να το πράξουμε αυτό θα έπρεπε να σκεφτούμε μία πολιτική ποιότητας που να μπορεί να χορηγήσει στους, στους παραγωγούς αυτών των προϊόντων ε, τρόπους να και εργαλεία να βελτιώσουν ε, τα προϊόντα και την παραγωγή τους, να υπάρξουν ε, κάποιες πολιτικές προγραμματισμού της παραγωγής και Επίσης κάποιες θεσμικές εκστρατείε για να προωθήσουν την αναγνωρισιμότητα όλων αυτών των σημάτων από τον καταναλωτή. Και τέλος να εξορθολογηθεί το σύστημα της πιστοποίησης για να είναι ε, και πιο αξιόπιστο σε διεθνές επίπεδο και να έχουμε προϊόντα που πραγματικά είναι διαφορετικά από τα υπόλοιπα προϊόντα που έχουμε στην αγορά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Παντίνη και τώρα καλούμε τον άλλο εμπειρογνώμονα, τον κύριο Ζιλελέφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την πρόσκληση στην παρουσίαση αυτή που αφορά την θέση των μικροκαλλιεργητών, το ρόλο των τοπικών αγορών στα γενικότερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ποιοτικής πολιτικής. Ε, θα αναφερθώ σύντομα στο γενικότερο πλαίσιο στο οποίο τίθεται αυτό το πρόβλημα. Τι λέει η δέσμη για την ποιότητα, ποια είναι η κατάσταση των μικρών αγροκτημάτων και μετά θα κάνω και μερικές συστάσεις. Για το γενικότερο πλαίσιο Θέλω να τονίσω συντομότατα και χωρίς να αναπτύξω μια αλλαγή που σημειώθηκε εδώ και 10-20 χρόνια στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το καθεστώς της ανταγωνιστικότητας διεθνώς. Στη δεκαετία του 90 είχαμε πει ότι υπήρξε στροφή προς τις υπηρεσίες ή την ποιότητα και δύο τάσεις σημειώθηκαν ως προς την ζήτηση των καταναλωτών και καταναλωτριών προϊόντα με νόημα που σώζουν τον πλανήτη κτλ. και ένα αίτημα για περισσότερες υπηρεσίες που περνούσε από εστιατόρια, συλλογική, συλλογικά, βιολογικά τρόφιμα κλπ. Στη γενικότερη αυτή αλλαγή θα ήθελα επίσης να σημειώσουμε μια αλλαγή του πολιτικού λόγου μετά την κρίση που οδηγεί στη διατύπωση ορισμένων ερωτημάτων όπως της διαχείρισης των συναλλαγών και της διευθέτησης μέσω της συμβατική οικονομία, οικονομία των συμβάσεων ή συμβολέων. Για την ποιοτική δέσμη έχουμε πει ότι ο αριθμός AUP και PGI αυξήθηκε από το 92, αλλά γενικότερα τα συστήματα εθελοντικής πιστοποίησης αυξήθηκαν 440 παριθμοί Κομισιόν και αφορούν και τη βιολογική γεωργία και τα ποιοτικά γενικώ προϊόντα. Επίσης, μεταξύ των καινούριων στοιχείων της δέσμης αυτής είναι ο ρόλος, η έμφαση που δίνεται στο ρόλο των ομαδοποιήσεων παραγωγών στη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών ποιοτική παραγωγής και αγορών. Η, τα μικροαγροκτήματα και τοπικές αγορές τώρα, από τη μία η δέσμη της ποιότητας τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι είναι δύσκολη η συμμετοχή των μικρών παραγωγών στα προγράμματα αυτά ποιότητος και από την άλλη η ανακοίνωση για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δείχνει τη σημασία που έχει η ποιοτική πολιτική μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανταγωνιστικότητας όχι μόνο προστασίας μερικών συστημάτων ή περιφερειών όπως στο παρελθόν αλλά ιδιαίτερα τονίζεται ο ρόλος του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας για την επανεξισορρόπηση των αγορών και ζητιέται η δημιουργία ενός συγκεκριμένου εργαλείου για τους μικροπαραγωγούς. Πρέπει να κάνουμε να διαχωρίσουμε εδώ την γεωργία μικρής, μικρών διαστάσεων με τη γεωργία για την επιβίωση η οποία παίζει ένα σημαντικό κοινωνικό ρόλο που εξαρτάται βέβαια από τη συγκυρία, από τη γενικότερη οικονομική συγκυρία ή από περιφερειακή συγκυρία και σημειώνεται ιδιαίτερα στις νέες χώρες μέλη, μόνο. Συνδέεται με μια άτυπη λειτουργία της οικονομίας και επίσης με την Εθνική Πολιτική Κοινωνικής Προστασίας. Και έχει μια πραγματική συμβολή στον αγροτικό κόσμο και στη βιοπικιλότητα. Η μικρών διαστάσεων γεωργία συμμετέχει στις τοπικές αγορές και ως προϊόντα και ως υπηρεσίες και χαρακτηρίζεται πρώτον από την αυτονομία της ως προς τα input και μπορεί κανείς να διαπιστώσει την εξέλιξη προς μεγαλύτερο αριθμό οικογενειακών και πρασίνων αγροκτημάτων Πράγμα το οποίο δεν αυξάνει μόνο τη βιοπικιλότητα αλλά και βοηθάει στην καλύτερη κατανομή της παραγωγής περιφερειακά, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές. Άρα χρειάζονται διαφορετικά μέτρα για τις διαφορετικούς αυτούς τύπους γεωργίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το καθεστώς του αγρότου και της αγροτήσης ε, δεν είναι απλώς αλλαγή του νομικού καθεστώτος που ήδη ισχύει. Η κατανομή των αγροκτημάτων ανάλογα με το μέγεθός τους διαφέρει όπως ξέρετε από χώρα σε χώρα της Ένωσης και αν σκεφτούμε μόνο τα μικρότατα αγροκτήματα δύο εκταρίων ή λιγότερο από δύο οικονομικών μονάδων αντιπροσωπεύουν παρόλα αυτά 44% του συνόλου των αγροκτημάτων ενώ μόλις 3% της επιφανίας. Τώρα, αυτό το 47% είναι στην πραγματικότητα χαμηλότερο, πολύ χαμηλότερο αν σκεφτούμε μόνο όσους ωφελούνται από τον πρώτο πυλώνα γιατί ανάλογα με τα όρια που έχουν τεθεί από την κάθε χώρα τα αγροκτήματα αυτά δεν έχουν πρόσβαση στην ουσία στον πρώτο πυλώνα. Αν δούμε τώρα όμως τα αγροκτήματα άνω των 10 εκταρίων πάρα πολλά παραμένουν μικρών διαστάσεων με οικογενειακή κυρίως εργασία. Η εφαρμογή ενός απλοποιημένου σχεδίου λοιπόν με αμέσων πληρωμών δεν απαιτεί καινούριο ορισμό των μικρών αγροκτημάτων. Γιατί υπάρχουν αγροκτήματα μικρά που θα έπρεπε να τύχουν κάποιας προσαρμογής και των μέτρων γενικότερα της ΚΑΠ παραδείγματος χάρη του δεύτερου πυλώνα και των μέτρων ποιότητος. Η γεωργία αυτή η επιβίωσης όπως λέω θέτει το πρόβλημα του ορίου εγγραφής ε, μετά το οποίο μπορεί κανείς να τύχει επιχορηγήσεων. Υπάρχουν αγροκτήματα που αυτή τη στιγμή αναπροσαρμόζουν τη λειτουργία τους Και από την άλλη μεριά για την μικρών διαστάσεων γεωργία υπάρχουν μηχανισμοί δικαιότερης κατανομής των πληρωμών από την ΚΑΠ παραδείγματο χάρη τα ανώτατα όρια αναεργαζόμενων για τις άμεσες πληρωμές ή η διατήρηση των ειδικών ταμείων με το απλοποιημένο σύστημα αμέσων πληρωμών αλλά υπάρχει και οικολογική διάσταση, η απλοποίηση των διαφόρων συστημάτων και των μηχανισμών που μπορούν να ενθαρρύνουν την μικρών διαστάσεων γεωργία. Το σημαντικό είναι και το δείχνουν ορισμένες μελέτες κυρίως στη Γαλλία αλλά και αλλού ότι αν η μικρών διαστάσεων γεωργία συμμετέχει λιγότερο από άλλων διαστάσεων γεωργία στα προγράμματα αυτά ποιότητας. Παρόλα αυτά το γεγονός παραμένει ότι και τα μικρά αγροκτήματα συμμετέχοντας σε αυτά τα προγράμματα αυξάνουν τις δυνατότητές τους επιβίωσης. Η βελτίωση της συμμετοχής της μικρής διαστάσεων γεωργίας στα ποιοτικά προγράμματα αφορά και υποδομές και συλλογικές επενδύσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Γενικότερα δεν απαιτεί περισσότερη πληροφόρηση για τα προγράμματα αυτά και μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύστημα διαβούλευσης. Στα πλαίσια μιας βιώσιμης ανάπτυξης, που να συμπεριλαμβάνει και την μικρών διαστάσεων γεωργίας, πρέπει, ε, γεωργία πρέπει να σκεφτούμε πρώτον την ανάγκη της διατήρησης των αποκτημάτων αυτών για τα τρόφιμα, για την παραγωγή τροφίμων και γενικότερα τα τροφιμικά συστήματα, πράγμα που μας οδηγεί να τονίσουμε πρώτον το ρόλο των περιφερειακών τοπικών προγραμμάτων που μπορούν να διευκολύνουν την ολοκλήρωση και των ε, περιβαλλοντολογικών υπηρεσιών αλλά και των ποιοτικών προγραμμάτων και από την άλλη το ρόλο των περιφερειακών προγραμμάτων στην μεγαλύτερη συνέπεια των παραγωγών για τρόφιμα. Οι επιπτώσεις των ποιοτικών προγραμμάτων θα ήθελα απλώ να πω τρία πράγματα μεταξύ όσων βλέπετε στην οθόνη. Ένα, ότι αυτά τα ποιοτικά προϊόντα, τα AUP ιδίως, διατηρούν ε, μια πολιτιστική κληρονομιά αλλά πρέπει και αυτά να προσαρμοστούν στις σύγχρονες αστικές μορφές κατανάλωσης. Σας έχω ήδη πει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για υπηρεσίες. Έπειτα, Μπορεί να δημιουργούν κοινά αγαθά και κοινωνικά και οικολογικά, αλλά αντιπροσωπεύουν ένα πρόβλημα για την ακριβή τους αξιολόγηση. Μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι οι ομάδες που παράγουν τέτοιου είδους ποιοτικά προϊόντα θα μπορούσαν όπως και οι μεγάλες επιχειρήσεις να κάνουν ένα είδους reporting στις δεσμεύσεις που μπορεί να αναλάβουν οικολογικά. Τονίζω ιδιαίτερα τον πολλαπλασιασμό των διαφόρων μαρκών και πιστοποιήσεων. Τώρα, για τα προβλήματα που έχουν οι μικρές εκμεταλλεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά, ας πούμε για το δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, Υπάρχουν και οικονομικοί φραγμοί ατομικοί που σχετίζονται με το κόστος εφαρμογής της πιστοποίησης και διανομής, αλλά υπάρχουν επίσης και πολιτιστικοί και κοινωνικοί φραγμοί. Πολιτιστικοί φραγμοί, δηλαδή τις πηγές της γνώσης και πληροφόρησης. Ο ρόλος των αγροτών με μικρές εκμεταλλεύσεις εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι πολλές φορές οι... υπάρχουν μεγάλες περιφερειακές εξαιρέσεις στην παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων. Καμιά φορά μιλάμε για το καλάθι περιφερειακών προϊόντων, ιδίως στις τουριστικές περιοχές. Αλλά και για νέες μορφές τοπικών αγορών για τις οποίες θα μιλήσω σε λίγο. Ξέχασα να σας πω πριν, να μιλήσω για τα προϊόντα του ποιοτικού συστήματος που είναι σημαντικά στις διεθνείς συναλλαγές αλλά ιδιαίτερα διανέμονται από τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές. Έχουν λοιπόν μεγάλη σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Άρα πρόκειται εδώ για αναγνώριση της σημασίας των λειτουργιών αυτών μέσω της συμμετοχής τους στην πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου. Τα υπόλοιπα της δέσμης ποιότητας αφορούν κυρίως την προσφορά, δηλαδή ήδη υπάρχουν, διαθέτουν πολλά μέσα ελέγχου της προσφοράς οι οικονομικοί παράγοντες και διαρθρωτικά μέσα όπως η τα όρια των ζωνών και γενικότερα τα αναπτυξιακά προγράμματα όσο μεγαλύτερη σύνδεση έχουν με τους τοπικούς πόρους τόσο περισσότερο μπορεί να ελεγχθεί η ποιότητα. Υπάρχουν όμως και άλλα μέσα όπως μια ιεράρχηση των τμήματων αγορών των προϊόντων αυτών όπως το κρασί αλλά μπορεί να ισχύει το ίδιο και για το τυρί και για το κρασί ας πούμε υπάρχει ένα σύστημα de facto ποσοστώσεων εμέσων μέσω του περιορισμού της παραγωγής ή των ορίων της παραγωγικότητας. Και υπάρχει βέβαια και το θέμα της αποθήκευσης αλλά ιδιαίτερα η δυνατότητα να δημιουργήσει κανείς δευτερογενείς αγορές, δηλαδή ένα τμήμα της παραγωγής του να το πουλά γενικώ ή με συγκεκριμένη μάρκα. Νομίζω ότι για τέτοιου είδους παραγωγή δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί ένα αυστηρό σύστημα ποσοστώσεων, αλλά παραμένει η αναγκαιότητα να προβλέπονται οι κρίσεις που μπορεί να πλήξουν τέτοιου είδους συστήματα παραγωγής. Και άρα, στην περίπτωση αυτή, ερχόμαστε στο θέμα της διευθέτησης της ενιαίας αγοράς και το ρόλο των συσσωματώσεων. Για τις τοπικές αγορές αυτές διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Ε, εδώ σημειώθηκε μια αλλαγή πρόσφαση πρόσφατες δεκαετίες. Δηλαδή έγιναν, γίνονται πωλήσει άτυπες ή οικογενειακές και τελευταία αναπτύχθηκαν και νέοι τύποι εναλλακτικοί Βλέπουμε τώρα ότι τέτοιου είδους προσπάθειες συνδυάζονται. Τα χαρακτηριστικά της νέας αυτής φάσης νομίζω ότι είναι τρία. Το ότι μερικοί γεωργοί χρησιμοποιούν αυτούς τους νέους τρόπους διανομής γιατί αντιδρούν έτσι τα προϊόντα χωρίς ετικέτα. Δεύτερον, λαμβάνουν υπόψη τους έτσι τη σημασία των υπηρεσιών στις νέες αυτές αγορές, όπως ας πούμε στη συλλογή, στα συλλογικά εστιατόρια ή στα μεγάλες αλυσίδες και γενικά στη διαχείριση της διατροφής. Τέλος, ορισμένες συστάσεις για, τις μικρών διαστάσεων, για τα μικρών διαστάσεων αγροκτήματα υπάρχει το θέμα των ε, βοηθειών επιχορηγήσεων για τις επενδύσεις ή πληρωμές ανά οικογένεια αλλά επίσης και η δυνατότητα συμμετοχής σε αγροπεριβαλλοντολογικά προγράμματα. Πώς όμως να δικαιολογήσει κανείς την απλοποίηση αυτών των ελέγχων, μία δυνατότητα θα ήταν, όχι με συγχωρείτε λάθος, για τα μικρά αγροκτήματα, όχι για τα που περι τα μικρά. Χρειάζεται βέβαια μια προσαρμογή στις ή των ατομικών, των ατομικών ε, συνηθιών, κάποια διοικητική στήριξη και καλύτερη πληροφόρηση, αλλά επίσης και κάποια χορήγηση βοήθειας των προγραμμάτων που έχουν σαφή περιφερειακή διάσταση. Όσο για τη συμμετοχή στα, σε οικολογικά προγράμματα των μικρών αγροκτημάτων θα μπορούσε κανείς να πει ότι δικαιολογείται Α, όχι, δεν εγώ δικαιολογείται, άραξα το... Δεν το... Λοιπόν. Ε, επανέρχομαι στα μικρά αγροκτήματα μία επιχορήγηση, μία στήριξη για την πιστοποίηση και μια αλλαγή στο σύστημα του ελέγχου. Αυτό εννοούσα ρε παιδί μου. Δηλαδή η συμμετοχή σε προγράμματα αγροτοπεριβαλλοντολογικά δικαιολογείται από τη συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα, προγράμματα ή σε συλλογικά προγράμματα με, με συλλογική ευθύνη. Γιατί πιστεύω ότι ως προς την ευθύνη πρέπει, δεν πρέπει να γνωρούμε ότι, ότι η χορήγηση κοινωνικών, κοινών αγαθών είναι κάτι συλλογικό, δεν αφορά ένα, ένα αγρόκτημα. Να, συλλογικό. Και είναι επίσης σημαντικό να υπάρξει εδώ μια συνέχιση τέτοιων δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο, όχι ατομικά περιφερειακό. Και θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε εδώ και στόχους κοινωνικής ολοκλήρωσης. Πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή λίγο τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι και οι αξιολογήσεις των με περισσότερη συλλογική ευθύνη και ίσως γιατί όχι και την δυνατότητα να χορηγηθούν περισσότερες στηρίξεις ή ένα τμήμα τους να βασίζεται στην επίτευξη μη των συλλογικών στόχων. Για τις κατευθυντήριες γαραμές και τα προγράμματα εθελοντικής πιστοποίησης που αναφέρονται πολλές φορές στα προβλήματα της βιώσιμης ανάπτυξης, μία σύστασή μου είναι να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία για τους οργανισμούς που καθορίζουν πρότυπα. Για την ανάπτυξη τοπικών αγορών βεβαίως πρέπει να ανταλλαχθούν εμπειρίες και καινοτομία, επιμόρφωση, υποδομές διαφοροποίηση των στηρίξεων αλλά και εδώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια αποτίμηση της συλλογική διάστασης των προγραμμάτων. Σας κατευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Κυρία Καρθία Περές. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους ε, δύο προηγούμενους ομιλητές για τη συνεισφορά του σε αυτό το σεμινάριο, για τις απόψεις που μας εκθέσανε που πιστεύω ότι μας ε, παρουσιάζουν ποια είναι η πρόκληση που έχουμε ονοποιών μας ε, πρώτης αναθεώρησης της δεσμής μέτρων για την ποιότητα. Νομίζω ότι τα στοιχεία που μας παρουσιάστηκαν μας δείχνουν ότι η ποιότητα των ε, ευρωπαϊκών διατροφικών προϊόντων ε, με σήμα ποιότητας ε, είναι μια προσθεμένη αξία, αλλά ακόμη δεν έχουμε μπορέσει να το μετατρέψουμε αυτό σε μια ευκαιρία σε διεθνές επίπεδο και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις πληροφορίες που δίνονται στον Ευρωπαίο πολίτη. Καταρχήν αυτή η Επιτροπή αντιμετώπισε θετικά τη δεσμή μέτρου που μας παρουσιάστηκε από την Κομισιόν. Αυτό σύμφωνα με όσα αρχικά λέγαμε για την έκθεση Σκότα. Εκεί είχαμε κάνει για κάποιες ενισφορές, κάποιες, είχαμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες, ορισμένες έχουν συμπεριληφθεί στην πρόταση της Κομισιόν, άλλες ε, έχουν μείνει εκτός, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα ξαναδούμε τα θέματα αυτά. Και καθώς δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα ήθελα να συμμετάσχουν στη ζήτηση και άλλοι συνάδελφοι, θα επικεντρωθώ σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα, επί των οποίων θα ήθελα να ακούσω ε, τους ομιλητές, γιατί αναφέρθηκαν στα θέματα αυτά. Ο κύριος Παντίνη μίλησε για το ρόλο του. Ε, ομάδων παραγωγών, αναφέρθηκε στον προγραμματισμό της παραγωγής. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε στον έλεγχο των όγκων παραγωγής. Είναι ένα θέμα επί του που εργαζόμαστε εμείς αυτή την Επιτροπή και βεβαίως ε, έχουμε δύο διαφορετικές ε, σκοπιές. Αφενός μιλάμε για προστασία δημόσια όπου οποιοδήποτε παραγωγός σέβεται τις προϋποθέσεις και έχει δικαίωμα ε, να παράξει βάσει της ονομασίας προέλευσης. Όμως είναι αλήθεια ότι αν κατά κάποιο τρόπο δεν είμαστε ικανοί να ελέγξουμε τους όγκους παραγωγής, μπορούμε, μπορεί να καταλήξουμε στις περιπτώσεις που μας εξέθεσε ο κ. Παντίνη. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τη γνώμη σας ακριβώς για αυτό το ζήτημα του ελέγχου του όγκου παραγωγής. Το έχουμε συζητήσει και το έχουμε παρουσιάσει και στην Κομισιόν και μάλλον είναι και μία από τις συζητήσεις που θα έχουμε επιτάπητος όταν θα συζητήσουμε το ίδιο τη δεσμή μέτρων. Και ένα άλλο ζήτημα που νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου είναι το εξή. Αυτή τη στιγμή στον κανονισμό για την ποιότητα και στον κανονισμό για τη θέση σε εμπορία στον κανονισμό ποιότητας, στο παράρτημα 2, έχουμε τώρα τις προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε για το ζήτημα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αν μιλάμε για ένα κανονισμό ποιότητας όπου θεσπίζονται κάποια πρότυπα, κάποιοι κανόνες που πρέπει να σέβονται και να πληρούν ε, η παραγωγή εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να διατηρηθούν σε αυτό τον κανονισμό ποιότητας οι διάφορες προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης στα κειμένα ειδικά προϊόντα και τα λοιπά και στη συνέχεια θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και τα ε, προϊόντα που προέρχονται από τις ειρηνές περιοχές και κατόπιν να αφήσουμε τις ε, γενικές ενδείξεις προαιρετικές ε, στους κανόνες για την εμπορία αν ε, ο στικό μα στόχο με την τροποποίηση των κανονισμών είναι να βελτιώσουμε την ενημέρωση που παρέχεται στον καταναλωτή, νομίζω ότι θα έπρεπε να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τι είναι ένα κανονισμό ποιότητα, όπω επιλαμβάνουμε ορισμένα προϊόντα που πληρούν ορισμένε προποθέσει αφενό και αφετέρου τον ίδιο τον κανονισμό εμπορία, όπου καθορίζονται τα πρότυπα που πρέπει να καθοριστούν. Οι κανόνε πρέπει να καθοριστούν. Δεν θέλω να με κρυγορήσω άλλο, συμφωνώ όμω, είπε ο κ. Παντίνη για τις κατεξουσιοδότηση πράξη. Νομίζω ότι με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Γνωρίζω ότι πρέπει να αναζητήσουμε αυτή την ισορροπία μεταξύ της ε, ταχύτητα. Ε, ε, ορισμένες έναντι ε, τις ε, θέσεις εφαρμογή ορισμένων πρωτοβουλειών, όμως υπάρχουν ορισμένα ζωτικά ζητήματα και φυσικά πρέπει να τοποθετείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ζητήματα αυτά και πρέπει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσει. Έτσι λοιπόν θα αναζητήσουμε με ισορροπία μεταξύ των κατεξουσιοδότηση πράξεων και των βασικών πράξεων όπου το Κοινοβούλιο μπορεί να γνωμοδοτήσει σχετικά. Αυτά σας ευχαριστώ. Are cuvântul în continuare domnul Dorfman. Καλώς συνεχίζονται κύριο Τόρφμαν. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι όσα ακούσαμε σήμερα το απόγευμα ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα Ήδη υπόθηκαν ε, από την προηγούμενο ομιλήτρια τα ουσιαστικά ζητήματα. Εγώ νομίζω ότι οι δύο προτάσεις Κομισιόν οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακόμη και αν ε, σήμερα τα αριθμητικά στοιχεία που μας παρουσίασε ο κ. Παντίνη δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Δηλαδή μόνο το 2% της ε, αξίας της αγροτικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τμήμα των προϊόντων με ένδειξη πρόληψης δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και βεβαίως θα πρέπει και να σκεφτούμε γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα του προγραμματισμού της παραγωγής είναι ζωτική σημασία. γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ το κατανοώ αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για ορισμένε ονομασίε ε, μια ονομασία είναι και η μάρκα. Κυρίω ε, στι μεγαλύτερε, στι διεθνεί αγορέ. Γιατί κανένας δεν μπορεί να μου πει ότι μια ονομασία όπως ε, το προσούτο από την Πάρμα, το ροκφόρ, η σαμπάνια δεν αποτελούν και ένα σήμα, μια μάρκα που πρέπει να τύχει αντικείμενο διαχείριση όπω ε, όλε οι υπόλοιπε μάρκε που έρχονται στην αγορά. Και το να διαχειριστούμε ένα σήμα σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσουμε πόσο εξ αυτού είναι στην αγορά. Και αν δεν δώσουμε αυτή τη δυνατότητα εμεί στου παραγωγού, δεν θα είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν επί του σήματο. Ε, επενδύουν επί της ιδιωτικής ε, μάρκας και όχι επί της ονομασίας προέλευσης. Εγώ είμαι ότι πρέπει να το σκεφτούμε το θέμα αυτό. Χωρίς να περιορίσουμε τους παραγωγούς, χωρίς να τους εμποδίσουμε να έχουν πρόσβαση στην αγορά των ονομασιών προέλευσης. πρέπει να ανοίξει μια δημόσια ονομασία σε όλους. Τώρα, για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, εδώ συμφωνώ με όσα υπόθηκαν. Θα πρέπει και εδώ να σταθούμε και να σκεφτούμε επί της πρότασης της Κομισιόν και να δούμε αν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται εκεί μπορούν πράγματι να επιληθούν με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. open πρέπει να σκεφτούμε κάπως πιο συγκεκριμένα θέματα. Σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι δυνατό ότι όλα όσο το μέσο της παραγωγής ε, θα περιοριστεί ε, στη ζώνη προέλευσης. Και εδώ αναφέρουμε και στην μεταποίηση, σε ποιο βαθμό είναι δυνατό μια κοινοπραξία, ένα consortium να αποφασίζει και για την ετοιμασία του προϊόντος στην λόγο περιοχή. Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο το θέμα της ε, ονομασίας προέλευσης για ε, ένα προϊόν που έχει τύχη επεξεργασίας. Ε, κοιτάξτε, εγώ τώρα να έχω ένα σάντουιτς και έχει μέσα ε, προσούτο από την Πάρμα μπορώ να γράψω προσούτο, ε, προσούτο από την Πάρμα δεν ξέρω αν είναι δυνατό να υπάρξει έλεγχος ίσως ναι αν δεν είναι δυνατό να υπάρχει ο έλεγχο, τότε δεν ωφελούμε κανένα, ούτε τον ε, παραγωγό, ούτε τον καταναλωτή, γιατί υπάρχει ο κίνδυνο ε, το προσούτο που θα καταλήξει στο σάντουιτς να μην προέρχεται τελικά από την πάρμα. πρέπει να σκεφτούμε και επί των ειδικών ενδείξεων για τις ορεινές περιοχές λόγου χάρη. Στο πρώτο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πρώτο σχέδιο κειμένου υπήρχαν και παραδόξως τώρα εξαφανίστηκαν. Και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε να επενεισαγάγουμε και το σήμα που προβλέπεται για ε, τα προϊόντα που ε, διανέμονται στις τοπικές αγορές. Αυτά είχα να πω, Πάντω θεωρώ ότι η δρόμο που ακολουθείτε είναι η σωστή. σα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ το λόγο έχει ο Ευχαριστώ. Με πολύ ενδιαφέρον παρακολούθησα τις δύο ε, ομιλίες. Ίσως λοιπόν να είναι μου να επικεντρωθώ λιγότερο στα στις ενδείξεις ποιότητας που παρόλα αυτά βέβαια και βλέποντας και πόσοι μίλησαν για το θέμα αυτό έχει κεντρική σημασία για την ε, ονομασία προελεύσεως και τις άλλες ονομασίες. Θα πρέπει λοιπόν οι οργανώσεις ε, που είναι αρμόδιες για την παραγωγή να είναι σε θέση να ελέγχουν ε, αυτά τα σημεία ποιότητας, αυτές, ε, τα χαρακτηριστικά ποιότητα για να μην χάσουμε τελείω όποια αξία μπορεί να έχει το σήμα ποιότητα. Ένα άλλο ζήτημα όμω είναι μεγάλο πρόβλημα για τα προϊόντα ονομασία προελεύσεω, οι απομιμήσει του. Όπου θα πρέπει να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτέ τι αγορέ, που σαν τον κούκο εγκαθίστανται στι αγορέ αυτών των προϊόντων προελεύσεω και τα που χωρίς κανέναν έλεγχο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά πάντως είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα αφήσεται και είναι σοβαρό. Μικρές εκμεταλλεύσεις. Έχω τρία ερωτήματα. Καταρχάς για την ε, διαφύλαξη των ε, μικρών ε, εκμεταλλεύσεων και την δυνατότητα ενδεχομένως δημιουργίας νέων μικρών εκμεταλλεύσεων. Ερωτώ λοιπόν αν υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την υποστήριξη των τοπικών αρχών στην στήριξη μέσων εργαλείων, νομοθετημάτων όπως αυτά που αφορούν ε, τις τοπικές αρχές και που θα επέτρεπαν στις μικρές αυτές εκμεταλλεύσεις να εξασφαλίσουν ε, είτε μια διαφορετική διέξοδο ε, είτε μέσα μεταποίησης, σε αγορά δηλαδή, μεταποίηση αυτών των προϊόντων. Και κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να συνεργαστούν οι τοπικές αρχές, οι φυστάμενες τοπικές αρχές ε, και δομές και οι δομές αυτές ε, των, των επιχειρήσεων, των εκμεταλλεύσεων. Επίσης, σε σχέση με, τα, με τις προδιαγραφές ποιότητας, Πρέπει να διαφοροποιούμε ανάμεσα στον βιομήχανο που μπορεί να παράγει 3 εκατομμύρια τόνους και ένα μικρό παραγωγό που μπορεί να έχει 50.000 κιλά, κιλά ή και λιγότερα. Ή μάλλον 50 κιλά ή και λιγότερα ε, την ημέρα. Άρα ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε σε θέση και να διακρίνουμε μεταξύ των αγορών, τοπική αγορά, περιφερειακή αγορά ή εθνική ή και διεθνής. Εδώ πρέπει να γίνει διαφοροποίηση. Διαφορετικά ούτε αγορά θα έχουμε, ούτε μικρές μεσές επιχειρήσεις θα έχουμε, ούτε μεταπίεση σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτά θέλω τη γνώμη σας. Και άλλο ένα ζήτημα της εγκατάστασης. Θα μου πείτε, δεν συμβαίνει συχνά, είναι μάλλον απίθανο ε, να γίνεται εγκατάσταση σε μικρές επιχειρήσεις. Και όμως είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε μικρές εκμεταλλεύσεις όπου ο κόσμος, ο νέος άνθρωπος έρχεται εσκεμμένα και επιλέγει να τοποθετήσει την επιχείρησή του. Φερρυπίν ε, για να κάνει ένα φούρνο που θα φτιάχνει ψωμί στην πινακωτή ή τυρί ή δύο-τρία πράγματα μαζί που θα προσφέρει στο πικέγωνα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το στηρίξουμε και μέσα από ένα πλαίσιο διαφορετικό, γιατί οι βοήθειε ενισχύσει του πρώτου πυλώνα δεν καλύπτονται τι ε, δυνατότητε, δεν προσφέρουν τι δυνατότητε στήριξη. Έτσι λοιπόν θα έλεγα, σε αυτή τη νέα ε, δυνατότητα ανάπτυξης της υπαίθρου δεν θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα κοιτάξουμε τώρα να ακούσουμε τις απαντήσεις των επιρρογνωμόνων μας με πρώτο τον κύριο Παντίνη. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που τέθησαν. που κυρίως έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό της παραγωγής. Προσωπική μου γνώμη λοιπόν είναι η εξή. Η αρμοπιθότητα θα ξεκινήσει υπογραμμίζοντα ε, τι ε, συνέπειε που μπορεί να έχουν αυτά τα συστήματα. Γιατί είναι διαφορετικά. Τα συστήματα παραγωγή αυτών προϊόντων απαρτίζονται από μια σειρά μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή, ε, η χαλιναγώγηση της παραγωγής έχει σαν αποτέλεσμα όλες οι ποσότητες που προκύπτουν από την παραγωγή αυτών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να καθιστούν ομοιόμορφα αυτά τα προϊόντα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο κίνδυνος αστάθειας των τιμών στην αγορά οδηγεί αυτά τα προϊόντα να είναι πιο παρόμοια με τη λογική της αγοράς. Δηλαδή γίνονται price taker. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν κατορθώσουμε να έχουμε μέσα προκειμένου να αποφύγουμε αυτές τις προβληματικές της αγοράς, ε, ε, τότε ένα, ένα από τα εργαλεία αυτά είναι δηλαδή ίδιος ο προγραμματισμός της παραγωγής, τότε διακινδυνεύουμε ο αντίκτυπος σε αυτούς τους μικρούς παραγωγούς να είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι σε κάποια άλλη επιχείρηση παραγωγής τροφίμων. Επίσης, το να έχουμε και παραγωγή που σχετίζεται με την επικράτεια, αυτό δεν σημαίνει ε, ότι ε, αυτός αποτελεί παράγοντα περσέ που περιορίζει ε, την παραγωγή. Έχουμε πάρα πολλά προϊόντα ε, για τα οποία υπάρχει μεγάλη δυνατότητα παραγωγής μεγαλύτερης ποσότητας. Επίσης, ο έλεγχο της παραγωγής δεν θα πρέπει να είναι ένας ε, αυστηρός, ε, περιοριστικός έλεγχος. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσει της αγοράς. Ε, τη στιγμή που βρίσκονται και άλλες διέξοδοι στο εξωτερικό παραδείγματος χάρη, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η αύξηση παραγωγής ή της εισόδου νέων παραγωγών στο σύστημα. Μια άλλη πτυχή που εθίγει από τον κύριο Ντόρφμαν ε, για τον έλεγχο των συστατικών ε, και για το ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο από τη στιγμή που υπάρχει πραγματική δυνατότητα ελέγχου. Θα μπορούσε να είναι ε, κατάλληλο, να είναι σκόπιμο να αναθέσουμε ε, στους ε, ομίλους, παραδείγματο χάρη στις οργανώσεις παραγωγών αυτή τη δυνατότητα να επιτρέπουν την δυνατότητα του σήματος POP για τα συστατικά τα προϊόντα. Πολλές φορές το τελικό προϊόν, το μεταπημένο προϊόν, αν φέρει αυτό το σήμα, έχει προσθεμένη αξία. Έτσι λοιπόν μπορεί να αποτελεί αυτό μια ίδια ευκαιρία να ε, μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό το σήμα και για τα τελικά προϊόντα. Euh, πιστεύω ότι όσον αφορά τη σημασία των προϊόντων ονομασία προελεύσεως. το ότι είναι πολύ περιορισμένο. Ναι, αλλά αυτό εξαρτάται και από τον τομέα. Φερρυπίνο, οι ίνοι δεν καλύπτονται ακόμη από τον κανονισμό. Στο πλαίσιο όμω της διεθνής αγοράς ίνου και κυρίως στην Ευρώπη, η κατηγοριοποίηση με βάση κάποια κριτήρια ποιότητας είναι ακριβώς αυτή που έχει σημασία και αποτελεί το μεγαλύτερο κουμερίδιο της αγοράς σχέση με τα μαζικής παραγωγής κρασιά που θεωρούνται δευτερεύουσες ποιότητας. Το ίδιο και στα τυριά. Άρα πρέπει να βλέπουμε το σύνολο και όχι μόνο κάποιους μεσού. Ως προς το θέμα των ελέγχων, των όγκων. Υπάρχει, πιστεύω, ένα διτό πρόβλημα. Αφενό με ένα έλεγχο του όκου, αφετέρου δε η κατανομή των αξιών μέσα στην αλήθεια δε εφόσον ποτέ αυτό μα ενδιαφέρει, ο μικρό παραγωγό. Για τον έλεγχο, προφανώ τέτοιου είδου προϊόντα ενέχουν αξία λόγω της κοινωνικής τους εικόνας, της, σημασία του σημασίας τους για την κοινωνία κτλ. Αλλά έχουν και αξία στην αγορά, λόγω περιορισμού της ποσότητας. Αγόρια αξία που ιδιορικά το είχε επισημάνει και έτσι δικαιολογούσε και τις τιμές των καλών ε, κρασιών. Έχει δηλαδή να κάνει με την ε, σπάνιδα του προϊόντος περισσότερο αυτή η αξία στην αγορά. Πάντως δεν νομίζω ότι μπορούμε έστω και με αυτά να βρούμε κάποια λύση γενική που θα μας επέτρεπε να περιορίσουμε τους ε, όγκους για τη στη λειτουργία τους και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την διαχείριση των συστημάτων και αγορών αυτών. Στις επιλογές τους υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία περιορίζουν την επιλογή με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται. Ίσως με την τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών να μπορούσαμε να ζητούμε και να ζητήσουμε επί τη ευκαιρία και την εξέταση των συνεπειών ως προς την αγορά αυτών των νέων τεχνικών όρων. Αλλά όπως υπόθηκε σημαντικό είναι και σε αυτή την ε, περίπτωση να δοθεί δυνατότητα για, τους, ε, ε, για τις ενώσεις των παραγωγών να συμμετάσχουν. Δεν νομίζω ότι είναι το θέμα τόσο, ότι μπορεί να έχει μια τόσο γενική λύση. Ή ότι πάντοτε η αξία θα κατανέμεται και πάλι υπέρ του μικρού παραγωγού. για τα ερωτηματικά που έθεσε ο κύριος Μποβέος προς τις μικρές επιχειρήσεις. Βεβαίως συμφωνώ μαζί του. Ίσως να συμπληρώσω κάτι στο υπόμνημά μας για το ρόλο των ε, τοπικών αρχών. Από, την, ε, από το χαμηλότερο από το κλιμάκιο μέχρι και την περιφέρεια. Για την ανάπτυξη ε, συλλογικών δομών, πράγμα το οποίο βλέπουμε να γίνεται και στη Γαλλία και την Ιταλία και τον Εμένο Βασίλειο. Βλέπουμε δηλαδή ε, παρεμβάσεις για την ανάπτυξη νέων αγορών, φερρυπίν, συλλογική εστίαση ε, και στις επιχειρήσεις και στα νοσοκομεία, μαζική εστίαση, ούτω καθεξής. Και έτσι ο ρόλος των τοπικών ε, αρχών σε περιφερειακό επίπεδο, τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τοπικών αγορών που επιτρέπουν την ανάληψη δράσεως και από νέους φορείς οι οποίοι είναι απαλλαγμένοι από τον ενδιάμεσο. Γιατί ξέρετε, παλιά είχαμε αυτού που λέγαμε αμαύς, που ναι, μεν είχαν σαν στόχο και τη διαφύλαξη μια κάποια ποιότητα, αλλά και την υποστήριξη του ε, καταναλωτή, ε, εδώ τώρα, του παραγωγού. Τώρα όμως έχουμε, ακόμη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, την, ε, έχουμε λοιπόν μεγάλη ζήτηση για προϊόντα τα οποία έχουν παραγωγή κοντά στο τόπο που θα καταναλωθούν. Υπάρχει αυτή η διέξοδος τώρα μαζί με την ανάπτυξη και την βιώσιμη ανάπτυξη επιδιώκουμε. Και αυτό σημαίνει ότι τη γεωργία πρέπει να δούμε και από την έποψη της ε, χρήστης ως μου, η παραγωγή μου. Άρα έχουν διτό ε, πλεονέκτημα τα τοπικά προϊόντα να προσφέρουν. Επίσης, έχουμε εξαιρέσεις ή παρεκκλήσεις σε διάφορα θέματα, ε, υγειονομικά για μια σειρά από κατηγορίες αγοράς και επίσης και στο πλαίσιο των τοπικών αγορών μπορούμε να εισαγάγουμε την έννοια της συλλογικής ευθύνης ή κάποιου τύπου έλεγχο ε, λιγότερο τυπικό και βραδύ, αυτό έλεγχο ενδεχομένω και παρεκκλήσεις που σχετίζονται με τα δεδομένα των τοπικών αγορών. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και πάλι τους δύο εμπειρογνώμονες μας και για τις παρουσιάσεις τους αλλά και για τις απαντήσεις που έδωσαν στους συναδέλφους. Τώρα, το σχέδιο έκθεση θα σταλεί για μετάφραση στις 21 Μαρτίου. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεση στις 11 και 12 Απριλίου και προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 3η Μαΐου. Mm. Και θέτησε στην Επιτροπή στις 20 Ιουνίου. Ε, η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 28 Μαρτίου στις 3. Σας ευχαριστώ.